Συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε. Έχουμε κάνει ήδη το ακαδημαϊκό τέταρτο. Ξέρουμε ότι είναι λίγο δύσκολο το πρωί. Λοιπόν, έχουμε ανταλλαγή απόψεων με την ομάδα των κουβανών που βραβεύτηκαν των κουβανών γυναικών. de Ντεμπλάνκο, γυναίκες στα άσπρα, από το 2010 βρεβεθήσεις με το βραβείο Ζαχάροφ σήμερα το πρωί έχουμε την ε, Έλενα Λαρίνγκα Λαρινάγα που τις εκπροσωπεί και τον Αλεχάνδρο Γκονσάλες Χάγα από το Πρατηρητήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Κούβα θα μας δώσουν ε, μία εικόνα, μία άποψη. Ο κύριος ε, Φαρίνιας δεν μπόρεσε να έρθει στην Ευρώπη λόγω του ότι δεν του εδόθη θεώρηση. Καταδικάσαμε ε, το γεγονός ότι δεν είχαμε δυνατότητα να τον συναντήσουμε. Και πιστεύω ότι είναι σημαντικό όταν οικοδομούμε γέφυρες με κάποιες γέφυρες να, τις, να τους επιτρέπουμε εν πάση περιπτώσει να συναντιούνται μαζί μας τουλάχιστον οι εκπρόσωποι τους. Ιδιαίτερα όταν μιλούμε για ανθρώπους που έχουν βρεβευθεί με το, βραβείο, με το βραβείο Σαχάροφ. Νομίζω ότι είναι ένα μήνυμα που πρέπει να διαβιβάσουμε η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου να μπορεί να συναντάται και να συζητεί για τα ζητήματα που αποσχαλούν τις ενεχόμενες χώρες. Η κυρία Λαρινάγα λοιπόν, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Και ευχαριστώ θερμά την Πρόεδρο. Κάποιοι από τους ε, ανθρώπους που βρίσκονται εδώ θα με θυμούνται γιατί εδώ και χρόνια υποστηρίζω την ομάδα των γυναικών στα άσπρα και ήθελα σήμερα να θέσουμε το θέμα των κοινωνικών συνθήκων ζωής των γυναικών στην Κούβα. Το καθεστώς ε, ασκεί περιορισμούς και πίεση σε οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα στην Κούβα. Εμείς ως γυναίκες στα άσπρα, ε, δημιουργήσαμε ένα δίκτυο γυναικών εκπροσωπώντας όλες τις γυναίκες που είχαν ε, υποβάλει καταγγελίες στην κυβέρνηση. Αντιληφθήκαμε ότι όλες οι γυναίκες στην Κουβά συμμερίζονται μια μεγάλη ανησυχία που είναι η βία κατά των γυναικών. που λαμβάνει χώρα όχι μόνο στα νοικοκυριά, ιδιωτικά, αλλά και δημόσια. Πέρυσι έγινε μια λεγόμενη θεωρητική συνταγματική μεταρρύθμιση που δεν αλλάξε και πολλά πράγματα. Θα αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο από το 20 έως το 28 με, με συγκεκριμένες συνταγματικές διατάξεις που συμπεριλαμβάνουν και τη βία κατά των γυναικών η οποία πλέον θα θεωρείται έγκλημα. Ήθελα να σας δώσω κάποια στοιχεία. Εγώ ζω στην Ισπανία. Κάνω μια σύγκριση μεταξύ της κατάστασης στην Ισπανία και στην Κούβα. Έχουμε 4.700.000 ενήλικες γυναίκες, 24 εκατομμύρια στην Ισπανία. Τα επίσημα στοιχεία στην Ισπανία Μιλούμε για 210 θανάτους μεταξύ του 2013 και του 2018. Δεν έχουμε επίσημα μεγεθή για την Κούβα. Α, για την αντίστοιχη χρονική περίοδο έχουμε, εν πάση περιπτώσει, καταφέρει να βρούμε 502 θανάτους να εντοπίσουμε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι επίσημα αυτά τα στοιχεία. Ήθελα λοιπόν εδώ στα πλαίσια της συμφωνίας που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει με την Κούβα να θέσει το θέμα αυτό. Μιλούμε για κοινωνική δικαιοσύνη, μιλούμε για την ε, δυνατότητα των γυναικών να συμμετέχουν στην ε, κοινωνική ζωή, στα κοινωνικά δρόμενα, να εκφράζουν την άποψή τους, να μην υφίστανται καταπίεση, να έχουν συνταγματική υποστήριξη γιατί πρόκειται για μια πατριαρχική κοινωνία η Κούβα και η ανεργία ή η αεργία των γυναικών θεωρείται απολύτως φυσιολογική στη χώρα αυτή. Μεταξύ άλλων. Και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό. Συμβαίνει λίγο πολύ σε πολλές χώρες, σε πολλές κοινωνίες αλλά σήμερα εγώ εδώ εκπροσωπώ τις γυναίκες που υποφέρουν όχι από όλα αυτά αλλά και από την πολιτική βία που καταγγέλουν τα κενά και τις ελλείψεις του καθεστώτος στην Κούβα. Ε, πολλές γυναίκες περιορίζονται στην, ε, στο σπίτι τους χωρίς να μπορούν να βγουν έξω και είναι κάτι σαν ε, κράτηση, κάτι σαν φυλάκιση κάποιου είδους, εχμαλωσία, εν πάση περιπτώσει. διότι όταν καταγγέλεις και ή ανήκει σε οποιοδήποτε δίκτυο, οργάνωση λοιπά, υποτίθεται από το καθεστώς ότι ε, έχεις προβήσει αντικυβερνητική, αντικρατική ε, ε, δράση και επομένως υφίστασε περιορισμούς, πρόστιμα, φυλάκιση λοιπά. Εμείς έχουμε παρουσιάσει τα, τα σχέδιά μας, τα προγράμματά μας για μια πραγματική συνταγματική μεταρρύθμιση, για ένα ανοιχτό σύστημα, για μια διαφάνεια. Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε. Ε, είναι σημαντικό το σώμα σας να συνεχίσει να ακούει αυτά τα πράγματα και να τα θέτει. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Αλεχάνδρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε Αυτή η δυνατότητα μας ε, επιτρέπει να επικαιροποιήσουμε την κατάσταση στην Κούβα. Το 2017, όπως όλοι γνωρίζουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κούβα έφτασαν σε μία συμφωνία συνεργασίας που επιτρέπει και μία γενικότερη αναθεώρηση κυβέρνηση της Κούβας όμως προέβη σε πολιτική καταστολής, όπως ε, το συνηθίζει. Τώρα δεν επιτρέπει την έξοδο από τη χώρα σε ακτιβιστές. Και η κυβέρνηση προβαίνει σε κατηγοριοποίηση των πολιτών τον οποίο δεν επιτρέπει την έξοδο από τη χώρα. Για παράδειγμα, ο Γκυγέρμο Φαρίνιας ήταν ένας από αυτούς που δεν μπόρεσε να βγει από τη χώρα για να βρεθεί εδώ μεταξύ μας σήμερα. Πολλοί είναι οι λόγοι για τους οποίους ζητάμε μία αναθεώρηση του πολιτικού διαλόγου μεταξύ Κούβας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δυστυχώς ε, δεν υπήρξε ένας εξορθολογισμός ε, του όλου πλαισίου. Η Κούβα δεν πέτρεψε την έξοδο 96 ατόμων, καθώς και 14 ακτιβιστών που θέλησαν να συμμετάσχουν σε διεθνείς δραστηριότητες. Πέντε από αυτούς θα έπρεπε να παρευρεθούν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταξύ των οποίων και ο Φαρίνιας. Επίσης, ο Χωσέ Ντανιέλ Φερέρ ήδη εδώ και πέντε μήνες βρίσκεται στη φυλακή με έγκλειστους του ποινικού δικαίου χωρίς καμία εγγύηση ότι θα βγει. Μπορεί να παραμείνει στη φυλακή ακόμα για ακόμα εννέα χρόνια. Δυστυχώς οι καταστολές ε, ενισχύονται ως προς τους ακτιβιστές που δεν μπορούν να φύγουν από τη χώρα. Αναφέρομαι σε αυτή την περίπτωση γιατί είναι πολύ κοντινή σε εμένα και δείχνει τη στάση των κουβανικών αρχών έναντι των πολιτικών ε, κρατουμένων. Πέρσι τον Οκτώβριο κυρώθηκε αυτή η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέθανε όμως μετά από 43 χρόνια στη φυλακή ο Ερνάντο Σούζα Φορτούνη, ο οποίος είχε δώσει πολλές και μεγάλες μάχες για τον εκδημοκρατισμό στην Κούβα. Δυστυχώς όμως ε, κλείστηκε στη φυλακή για 43 χρόνια και φυσικά έχασε και τη ζωή του. Αυτό μας λυπεί ιδιαίτερα, διότι είχα την τιμή να βρεθώ να είμαι συγκρατούμενος με αυτόν τον άνθρωπο για πολλά χρόνια θα θέλαμε να προβούμε σε ορισμένες συστάσεις που θα έπρεπε να ενσωματωθούν σε αυτή τη συμφωνία εάν θέλουμε πραγματικά να ευεργετηθούν οι πολίτες της Κούβας. Σε... Πρώτον, σε σχέση με, τις, ε, με τα είδη συμφωνηθέντα, πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει μία διαδικασία κύρωσης των διεθνών συμφωνιών στον τομέα των πολιτικών, κοινωνικών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να μην είναι κάτι το προαιρετικό. Επίσης θα πρέπει να ενσωματωθεί η παραγραφή των διακρίσεων για πολιτικούς λόγους και να μην υπάρχουν ποινικέ και διοικητικές κυρώσεις κατά πολιτών για δραστηριότητες, για κοινωνικές και πολιτικές δραστηριότητες και να, επίσης να αποφυλακιστούν όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι. Επίσης, η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να μπορέσει να συμμετάσχει στον πολιτικό διάλογο, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει μέχρι τώρα. Θα πρέπει να προβλεφθεί ένας μηχανισμός διαλόγου όπου θα μπορέσουμε να υπερασπιστούμε τις αρχές μιας δημοκρατικής Κούβας. Επίσης, χρειάζεται ένας μόνιμος μηχανισμός έτσι ώστε οι πολίτες να μπορέσουν να προσφύγουν κατά των κρατικών αρχών όταν γίνονται παραβιάσεις ανθρωπίνων και δημοκρατικών δικαιωμάτων. Όσο προς το κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, η συμφωνία θα έπρεπε να επιβάλλει την ε, εφαρμογή των αρχών του ΔΟΕ και να μην υπάρχει αφαίρεση ή παρακράτηση μισθών όπως γίνεται από τις ε, κουβανικές αρχές μέσα στα πλαίσια των ε, εξωτερικών επενδύσεων. Ως προς τις επιχειρήσεις, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα πρέπει να εφαρμόζουν τις, έβγες, τις ίδιες εργασιακές και δεοντολογικές αρχές, ιδιαίτερα ως προς τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν δημόσια επιδότηση. Η συμφωνία θα πρέπει να απαγορεύσει τις διακρίσεις ως προς την είσοδο και έξοδο από τη χώρα των κουβανών πολιτών. Στο διαδικαστικό τομέα αυτής της συμφωνίας θεωρούμε ότι θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή μία ιεράρχηση έτσι ώστε να υπάρχει μία μεταβατική φάση για τους διάφορους τομείς συνεργασίας συνεργασίας οικονομικής και κοινωνικής φύσης μέχρι ότου αποδειχτεί ότι οι κουβανικές αρχές τηρούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και καταβάλουν δίκαια τους μισθούς. Σε σχέση με ε, τις δημοκρατικές αρχές θα πρέπει να υπάρχει μία ειδική ρήτρα υπέρ των δημοκρατικών αρχών έτσι ώστε να μπορέσει να καταγγελθεί η συμφωνία εάν παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το κουβανικό παρατηρητήριο είναι πεπισμένο ότι κάτι τέτοιο δεν θα γινόταν αποδεκτό, ένα τέτοιο καθεστώς δεν θα γινόταν αποδεκτό από καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει λοιπόν να μη ληφθεί υπόψη αυτό το πλαίσιο ιδιαίτερα ως προς μια στρατηγική συμφωνία και όπως βλέπουμε ότι ισχύει ως προς τις εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ. Αυτό αφορά ένα μηχανισμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς να κινηθούμε σε μία εθελούσια βάση. Γιατί αυτό δεοντολογικά δεν θα ήταν αποδεκτό. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, υποστηρίζω τις συστάσεις, τις συστάσεις σας και όλες αυτές οι συστάσεις βεβαίως δεν μας βρίσκουν όλους σύμφωνους. Δυστυχώς, όταν ψηφίζουμε στην Ολομέλεια, βλέπουμε ότι οι συστάσεις της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν την χάνουν συμφωνίας από άλλες χώρες ή κομμουνιστικά καθεστώτα, οι χώρες που υποστηρίζουν κομμουνιστικά καθεστώτα. Και γι' αυτό ε, θεωρώ ότι το δικό σας μήνυμα θα εισακουστεί στην Ολομέλεια, αλλά όχι από όλους, δυστυχώς. Η κυρία Βίσλερ έχει το λόγο. Ναι, ευχαριστήσω θερμά τους ε, δύο ομιλητές για τις μαρτυρίες τους. Εμείς πρέπει να πω ότι προσπαθούμε, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να υποστηρίξουμε τις οργανώσεις γυναικών όπου οι γυναίκες βρίσκονται υποκαταπίεση. Σίγουρα μπορείτε να υπολογίζετε στην υποστήριξή μας εκεί που μπορούμε να την ε, δώσουμε, να την προσφέρουμε. Ε, άκουσα με μεγάλη προσοχή τον κύριο Χάγα άκουσα τις συστάσεις σας οι οποίες ε, μου είναι πολύ γνώριμες διότι ανεξαρτήτως της χώρας για την οποία συζητούμε η τελευταίο, το τελευταίο ψήφισμα που είχαμε ήταν για το Βιετνάμ όλα αυτά που μας συστήνεται είναι αυτά που ζητούμε και εμείς ακριβώς το τελευταίο ψήφισμα που εγκρίναμε και ελπίζω πραγματικά να μπορέσουμε να κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή και ένα από τα πιο επίγοντα ζητήματα που ελπίζω πραγματικά να μπορέσει να υλοποιηθεί από την Επιτροπή είναι αυτές οι οργανωμένες καταγγελίες των πολιτών από ανεξάρτητο φορέα κάτι ελπίζω που θα μπορέσουμε να οργανώσουμε και στην Κούβα να συστήσουμε και σε άλλες χώρες με τις οποίες έχουμε συμφωνία σε Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλω τώρα να μακρηγορήσω και να στερήσω το λόγο από άλλους συναδέλφους, αλλά όλα αυτά τα ζητήματα που αναφέρατε και για το χρονοδιάγραμμα, ότι πρέπει να είναι σαφή αυτά που ζητούμε, με πολύ συγκεκριμένες χρονικές περιόδους βημάτων, γιατί δεν το ζητούμε απλώς εμείς. Ε, πρόκειται για μια συμφωνία που το άλλο μέρος της δεσμεύεται. Δηλαδή δεν είναι ότι επιβάλλουμε εδώ αν θέλετε κανόνες ευρωπαϊκούς αλλά είναι κανόνες που συμφωνούμε από κοινού. Και νομίζω ότι υπό την αυτή δεν είναι αδύνατον να επιτύχουμε κάτι. Προτού δώσω το λόγο σε κάποιον άλλον. Όπως είπατε είναι απολύτως απαράδεκτο ο άνθρωπος που είχαμε προσκαλέσει να μην μπόρεσε να έρθει, να, μην μπόρεσε να βγει από τη χώρα. Αλλά ακριβώς αυτή είναι η φύση και τα μέσα που χρησιμοποιεί το καθεστώς αυτό για όσους χρειάζονται περαιτέρω αποδείξεις δηλαδή. Έχουμε πλέον λοιπόν ένα απτό παράδειγμα μη συνεργασίας. Εμείς θα εξακολουθήσουμε να ζητούμε να υπάρξουν αποστολέ επισκέψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κούβα και αν υπάρξει άρνηση θα είναι και αυτό ένα προηγούμενο. Σα ευχαριστώ και πάλι και ελπίζω να μπορέσουμε σύντομα να έχουμε ένα μηχανισμό υποβολής καταγγελιών ανεξάρτητο. Για όσους διώκονται. Ώστε αυτοί να μπορούν να έχουν έναν συνομιλητή. Σας ευχαριστώ πολύ. Για τους σοσιαλιστές, ο Νάτσο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ την ε, κυρία Λένα και τον ε, Αλεχάνδρο και εγώ πολύ λυπούμε που δεν μπόρεσε να είναι εδώ ο κύριος Φαρίνιας που είχαμε προσκαλέσει του στέρισαν δηλαδή την θεώρηση που είχε ζητήσει και η Ισπανική Πρεσβεία μεταξύ άλλων. και είναι λυπηρό που δεν έχουμε φωνές που εκπροσωπούν την ε, κοινωνία στην Κούβα. το οποίο είχαμε τιμήσει και με τη βράβευσή του για το κοινωνικό του έργο. Παρότι δεν συμφωνούμε ε, σε όλα τα ζητήματα, όπως είπε και η κυρία Αρένα για τον Φερέρ, είχαμε ζητήσει την απελευθέρωσή του σε πλαίσια πιο ανθρωπιστικά παρά πολιτικής δηλαδή απέτησης. Επαναλαμβάνω έχοντας διαφορές. Εμείς υπερασπιζόμαστε τα πλαίσια, το πλαίσιο της συμφωνίας του πολιτικού διαλόγου με την Κούβα και όπως έλεγε η πρόεδρος επαναλαμβάνω δεν συμφωνούμε όλοι σε αυτό εδώ το κοινοβούλιο ή στο πλαίσιο αυτό, αλλά λέμε γιατί απλό. 20 χρόνια κυρώσεων δεν έχουν βοηθήσει κανέναν. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει άλλες λύσεις για να μπορέσουμε να καταφέρουμε βελτιώσεις πρόοδο που 20 χρόνια ε, αυστηρότατης και υπερήφανης στάσης ε, που τήρησε η Ευρωπαϊκή Ένωση υπό την καθοδήγηση του κυρίου Αθνάρ δεν οδήγησαν πουθενά και σε τίποτα. Πρέπει να βρούμε μια άλλη λύση. Ήθελα να ευχαριστήσω και τους δύο μιλητές και άλλους που είχαμε δει πρόσφατα για την ε, ευελιξία τους, πώς να το πω, δεχόμενοι ότι δεν μπορούν να πετύχουν τα πάντα, θυσιάζοντας δηλαδή μερικά από τα σημαντικότερα αιτήματά τους, ε, προσπαθούν να σημειωθεί μια πραγματική πρόοδος, να ζητήσουν σιγά σιγά απλά πράγματα. Και νομίζω ότι από την κουβανική αντιπολίτευση από τους αντιφρονούντες ε, με μια τέτοια στάση θα μπορούσαν να επιτευχθούν κάποιες βελτιώσεις. Κάποιες πραγματικές πρόοδοι. Και αν ε, συνδυάσουμε στο πλαίσιο της συμφωνίας ένα αίτημα με κάτι άλλο, ε, χωρίς να αρνούμαστε τον πολιτικό διάλογο, η δική μας η ομάδα σίγουρα είναι διατεθειμένη να το υποστηρίξει αυτό. Η δημοκρατική ρήτρα είναι, αν θέλετε, η πυρηνική διάταξη της συμφωνίας. Και ακριβώς επειδή είδαμε ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαμε πετύχει τίποτα, είμαστε πολύ... Ε, έχουμε μεγάλες αμφιβολίες για να ενεργοποιήσουμε αυτή τη ρήτρα. Πρέπει να κατανοήσει το καθεστώς στην Κούβα ότι η εικόνα που έχει πλέον προς τα έξω, η ιδεολογική του στάση να θέλει να δημιουργήσει μια ιδεώδη κοινωνία είναι ουτοπία. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υφίσταται και πολλές κοινωνίες προχωρημένες όπως είναι οι ευρωπαϊκές έχουν πολλά προβλήματα. Έχουν πολλά προβλήματα ισότητας των φύλων. Πώς να σκεφτεί κανείς ότι μια χώρα ε, με μια πατριαρχική παράδοση ε, δεν θα έχει τέτοια προβλήματα. Αλλά πάντοτε προσπαθεί το καθεστώς η κυβέρνηση της Κούβας να δώσει μια ιδεώδη εικόνα των πραγμάτων και εμείς προφανώς δεν μπορούμε να διδεχθούμε. Είναι σημαντικό λοιπόν η αντιπολίτευση στην Κούβα να, μην, να τοποθετείται όσο πιο ελεύθερα γίνεται. Και εδώ ακριβώς αυτά είναι τα κενά και οι ελλείψεις ε, του συστήματος κοινωνικής προστασίας στην Κούβα. Δηλαδή οι κοινωνικές ελευθερίες, τα αιτήματα των πολιτών εφόσον δεν υπάρχει κάποιος νόμος ή κάποια διάταξη που λέγει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν ή ότι δεν μπορούν να υπάρχουν κοινωνικές ελευθερίες, συγκεκριμένα και αυτά αιτήματα μπορούν ίσως να υποβληθούν σε ένα επίπεδο και αυτή η προσέγγιση που πολλοί είχαμε στο παρελθόν ότι πρώτα πρέπει να αλλάξουν τα οικονομικά πράγματα και μετά θα έρθουν όλα τα άλλα ε, έχει αποδειχθεί απολύτως λανθασμένη. Τα είχαμε δει και στο παρελθόν στο ψυχρό πόλεμο με τη Σοβιετική Ένωση. Ε, πρέπει να μην μετατραπεί όλο αυτό το, το πλαίσιο σε μια μετοπική αντιπαράθεση. Να μιλούμε για συγκεκριμένες κοινωνικές ελευθερίες, για, για την βία κατά των γυναικών. Τι κάνει η Κούβα, η κυβέρνηση της Κούβας, ε, δηλαδή υπάρχει κάποιος, κάποιο ιδεολογικό πρόβλημα βάσει του οποίου η κυβέρνηση της Κούβας δεν μπορεί να προστατεύσει τις γυναίκες της χώρας λόγω κάποιας πατριαρχικής πατροπαράδοτης αξίας. Δεν νομίζω ότι συνάδει με την ιδεολογία τους αυτή είναι η συνταγή που πρέπει να ακολουθήσουμε, να χρησιμοποιήσουμε το πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου που έχουμε θεσπίσει. Αυτό πρέπει να το μετατρέψουμε σε ένα πεδίο απαιτήσεων ε, εν είδη διαλόγου. Απαιτήσεων όμως. ενσωματώνοντας ε, μηχανισμούς ε, παρακολούθησης, παρατήρησης, αξιολόγησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα. Και είναι επίσης σημαντικό να έχουμε φωνές που να μην είναι μόνο αποκλειστικώς συνδεδεμένες με τους αντιφρονούντες ή με την ε, οργανωμένη αντιπολίτευση. Ε, ζητώ συγγνώμη πρόεδρε γιατί μακρηγόρησα. Ε, πάντως εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ τους δύο μιλητές. Αυτός, αυτό είναι το πολιτικό πλαίσιο που θεωρούμε ότι είναι κατάλληλο. Είναι ε, πλαίσιο εντός του οποίου μπορούμε να παρουσιάσουμε τις απαιτήσει μας, να συζητήσουμε και ίσως να οδηγηθούμε σε μικρές βελτιώσεις του κοινωνικού πλαισίου. Η κυρία Ροντρίγκε, παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για τις παρεμβάσεις σας και καταρχήν θα ήθελα να καταγγείλω. Λυπάμαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι ο κύριος Φαρίνιας δεν μπόρεσε να παρευρεθεί εδώ σήμερα. Ε, είναι λυπηρό και νομίζω ότι το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας θα πρέπει να καταδικάσει αυτή την πράξη και όπως είπε και ο ε, προλαλής σας, δεν ε, το απαγορεύτηκε μόνο η έξοδος, αλλά τελεί υποκράτηση. Πρόκειται για στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων στην Κούβα. Άλλη μια περίτρανη απόδειξη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ε, για την θεώρησή σας σήμερα. Μιλάτε για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία δυστυχώς ε, δεν τηρούνται. Ιδιαίτερα όταν οι γυναίκες ε, είναι πιο ευάλωτες και υφίστανται διακρίσεις στη Λατινική Αμερική αλλά και στην Κούβα. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό σήμερα είναι να δούμε αυτή τη θεώρηση πραγμάτων στην Επιτροπή μας, διότι σε όλα τα καθεστώτα όπου δεν υπάρχει ένα δημοκρατικό σύστημα ελεύθερης έκφρασης και αναγνώρισης πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, Φυσικά αυτές που πλήττονται περισσότερο είναι οι πιο ευάλωτες κατηγορίες, δηλαδή γυναίκες και τα παιδιά. Διότι χωρίς πολιτικά και δημοκρατικά δικαιώματα, τότε βρισκόμαστε ενώπιον μιας χώρας όπου δυστυχώς παραβιάζονται τα δικαιώματα κυρίως των γυναικών μέσα στα πλαίσια των διακρίσεων μεταξύ των δύο φύλων. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ότι υπάρχουν θετικές διακρίσεις πολλές φορές, αλλά στην προκειμένη περίπτωση στις ε, γυναίκες σε αυτό το νησί βλέπουμε, βλέπουμε ότι οι γυναίκες αποτελούν αντικείμενο μάλλον διακρίσεων, σοβαρών διακρίσεων. Θα πρέπει να δούμε τα πράγματα υπό αυτό το πρίσμα, διότι όπως είπε και ο Νάτσο, πολλά χρόνια περιμένουμε και τώρα θα πρέπει να απαιτήσουμε αλλαγές. Ουσιαστικές αλλαγές, γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε απαιτητικοί και ακέραιοι στις επικρίσεις μας για να μπορέσουν να γίνουν μερικά βήματα στην δημοκρατική διαδικασία. Αυτό που ζούμε σήμερα σε αυτή την Επιτροπή με την απουσία του κυρίου Φαρίνιας τα λέει όλα. Γιατί όπως ε, ξέρετε του χορηγήθηκε το βραβείο Ζαχάροφ το 2010 και αυτό δείχνει πολύ περισσότερο πολύ περισσότερα από οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό με λυπεί ιδιαίτερα η απουσία του. Σας ευχαριστώ πολύ για την δική σας παρουσίαση. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχουν άλλες ε, παρεμβάσεις. Ναι, έχετε το λόγο. Ιζαμπέλ. Δεν θα ήθελα να παρέμβω εξ αρχής, αλλά δεν μπορώ να μην το κάνω μετά από όλα αυτά δεν μπορούμε απλώς να αναφερόμαστε σε απουσίες, στην απουσία του κυρίου Φαρίνιας. Χρειάζεται δράση και νομίζω ότι η πρόεδρός μας θα πρέπει να αναφερθεί σε αυτές για να υπάρξει πραγματικός διάλογος μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κούβας θα πρέπει να αναφερθούμε και στα αρνητικά, διότι όλα αυτά ε, φέρουν και ένα μήνυμα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μόνο, όχι μόνο ο κύριος ε, Φαρίνιας δεν μπόρεσε να βγει από τη χώρα του, αλλά τελεί υποκράτηση. Δεν μπορούμε να πούμε όταν πρόκειται για δικτατορικά καθεστώτα ότι είναι πιο συμπαθητικά ή λιγότερο συμπαθητικά. Οι δικτατορίες είτε της δεξιάς είτε της αριστεράς είναι οι ίδιες. Το γεγονός ότι απαγορεύεται σε κάποιον να εκφραστεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ένα γεγονός το οποίο θα πρέπει να επιτείνει τη δράση μας. Θα πρέπει να γίνουμε ακόμα πιο απαιτητικοί αν πιστεύουμε στην Ευρώπη, σε μια Ευρώπη των αξιών, των δημοκρατικών αξιών. Είτε μιλάμε για πολιτικές ή εμπορικές σχέσεις, όλες αυτές θα πρέπει να υπόκεινται σε συγκεκριμένες αρχές. Και αυτό έχει σχέση με μεμονωμένες χώρες ή με μπλοκ χωρών. Το γεγονός ότι δεν γίνεται πυρηνική έκρη, έκρηξη με βάση ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να δράσουμε. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο εμείς έχουμε αρχές και υπεραμεινόμαστε των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αν δεν θέλουμε να πατήσουμε το κουμπί, τουλάχιστον θα πρέπει να αποστείλουμε σαφή μηνύματα από την Επιτροπή μας. γιατί έπονται και άλλες συμφωνίες στην ευρύτερη περιοχή της Λατινικής Αμερικής και θα πρέπει να γνωρίζουμε πού και πώς θα επιμείνουμε σε ένα παρόμοιο διάλογο. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω κατά πόσο έχετε κάτι άλλο να αναφέρετε εσείς. Σε σχέση με τις συστάσεις σας θα είχα να πω κι εγώ κάτι άλλο. Αναφέρεστε σε ένα μηχανισμό κυρώσεων, κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντί χωρών όπως η Κούβα, ένα μηχανισμό καταγγελιών, την εφαρμογή του εργασιακού δικαίου έχετε προβάλει αρκετές συστάσεις. Πιστεύετε ότι εάν οι συστάσεις αυτές δεν ενσωματωθούν στην εμπορική συμφωνία, θα πρέπει παρόλα αυτά να υπογραφεί η συμφωνία. Θέλω τη γνώμη σας, διότι πολλές φορές ε, λέμε ας ε, κυρώσουμε τις εμπορικές συμφωνίες και μετά θα δούμε. Όμως, ίσως θα πρέπει να είμαστε πιο απαιτητικοί για να φτάσουμε στους στόχους μας. Στην περίπτωση της Κούβας, τι πιστεύετε εσείς ως εκπρόσωπος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μετά από 20 χρόνια διαλόγου με τη χώρα αυτή. Πρόεδρε, πράγματι θεωρούμε ότι θα ήταν σφάλμα να μην ενσωματωθούν αυτές οι απαιτήσεις αυτές οι διατάξεις. Εμείς αυτό ζητούσαμε και συνοδεύσαμε όλη αυτή τη συζήτηση των προηγουμένων ετών, προτού κλείσει δηλαδή η συμφωνία, με αυτό το ίδιο αίτημα. Εάν αυτά τα στοιχεία δεν ε, ε, ενσωματώθηκαν ήδη στην συμφωνία δεν ήταν επειδή εμείς δεν το ζητούσαμε, το ζητούσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Υπήρξε μία στάση διευκόλυνσης προς την ε, κουβανική κυβέρνηση αλλά ακριβώς λόγω του ανοίγματο αυτού θεωρούμε ότι θα έπρεπε να είναι προαπαιτήσεις αυτές προκειμένου να υπογραφεί η συμφωνία. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι έχουμε εκπρόσωπο της πρεσβείας της Κούβας. Δύο λεπτά να τον ακούσουμε και μετά την ΙΕΒ παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω την ευκαιρία αυτή. Ε, νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να έχει μια ευρύτερη εικόνα, να ακούει περισσότερες φωνές, να ακούει πραγματικούς εκπροσώπους της κουβανικής ε, κοινωνίας, ε, όλους αυτούς που μάχονται για μια καλύτερη κοινωνία, αντί να προσκαλεί διαρκώς τις ίδιες οργανώσεις, τους ίδιους εκπροσώπους, τους ίδιους ανθρώπους, γιατί παρότι μπορεί να έχουν μια βράβευση Ζαχαρόφ, δεν έχουν κοινωνική στήριξη στην Κούβα. γιατί ε, κανένας από αυτούς ε, δεν μπόρεσε να εκλεγεί στο, στο παραμικρή, στην παραμικρή θέση κανένας εκπρόσωπος αυτών των μικρών ομάδων. Θα ήταν ενδιαφέρον να μας εξηγήσουν αυτοί οι κύριοι πώς είναι δυνατόν να αυτοαποκαλούνται οι υπερασπιστές των ε, ανθρωπιών δικαιωμάτων όταν απαιτούν την, τον οικονομικό αποκλεισμό και τις κυρώσεις που επιβάλλουν οι Ηνωμένε Πολιτείε οι οποίες εμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας και καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των γυναικών στη χώρα. Εγώ θα ήθελα να θυμίσω ε, τα κεφάλαια 3 και 4 της συμφωνίας που ακριβώς αφορούν ε, στην ευημερία των ε, πολιτών και των επιχειρήσεων και θα έπρεπε να είναι αντικείμενο εξέτασης από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, νομίζω ότι οι νίκες του λαού μας κατά τον παρά τις που έχουν επιβάλει οι Αμερικανοί, οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι ε, χαρακτηριστικές. Επίσης θα ήθελα να πω ότι ε, οι κρατήσεις στην Κούβα δεν γίνονται ε, έτσι όπως τις περιγράφετε εσείς, ε, ακολουθούν το δικαστικό, τις δικαστικές ε, αποφάσεις και διαταγές, γίνονται σύμφωνα με τα όσα ε, διατάσσει το δικαστήριο και δεν γίνονται απλώς ώστε να περιοριστεί ο λόγος ή η ελευθερία των απόψεων συγκεκριμένων οργανώσεων σε πολλές περιπτώσεις από αυτές τις οργανώσεις ε, ε, μιλούμε για εκπροσώπους ε, στην ουσία ξένων συμφερόντων και κυρίως αμερικανικών. Ως προς την περιορισμό της, ελε... ελευθερίας εξόδου οι αρμόδιες αρχές μπορούν να στερήσουν από συγκεκριμένο πολίτη την θεώρηση όταν υπάρχουν συγκεκριμένες δικαστικές αποφάσεις. όταν μιλάτε για τα δικαιώματα των γυναικών και καθότι σε καμία χώρα δεν έχουμε ε, ιδεώδες ε, συνθήκες ε, διαβίωσης των γυναικών, νομίζω ότι όταν οι γυναίκες στο παρελθόν περιορίζονταν στον νοικοκυριό και δεν είχαν καμία άλλη δυνατότητα, εντός του πλαισίου της Επανάστασης στην Κούβα σημείωσαν πραγματικές πρόοδου. Νομίζω ότι το προσδόκιμο ζωής ήδη των γυναικών έχει βελτιωθεί τόσο πολύ στην Κούβα που δείχνει την καλύτερη διαβίωσή τους. Είναι 60% των επαγγελματιών ε, της υγείας και της επαιδείας νομίζω στη χώρα μας, αν ακούσαμε καλά την ομιλήτρια, η οποία διαβάζει πάρα πολύ γρήγορα δυστυχώς. Ε, η πρόεδρος διακόπτη, δεν ακούμε την ομιλήτρια. Νομίζω ότι συνεχίζει η ομιλήτρια, όλες οι γυναίκες στην Κούβα έχουν ε, δικαίωμα ίσου μισθού για ίση εργασία. Η πρόεδρος όμως διακόπτει και λέει, θα... κοιτάξτε δεν γίνεται, δεν έχετε άλλο χρόνο. Είχατε το λόγο ως εκπρόσωπος της πρεσβεία της Κούβας, το οποίο δείχνει ότι έχουμε ένα πνεύμα διαλόγου με την ε, Κούβα. Εγώ λυπούμε και το λέω ως πρόεδρος της υποεπιτροπής ότι δεν είχαμε εδώ τους ανθρώπους που είχαμε προσκαλέσει προκειμένου να έχουμε έναν γαλήνιο διάλογο συζήτηση για το όσα συμβαίνουν στη χώρα σας. Ακούσαμε την τοποθέτησή σας. Ε, είναι σημαντικό ότι για την επόμενη ε, έκθεση που θα έχουμε ε, στον, στα πλαίσια του διαλόγου με την Κούβα για τα δικαιώματα του ανθρώπου και την ελευθερία έκφρασης να είναι προτεραιότητα αυτό και για εσάς και να έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε όλους αυτούς που κατά την άποψή μας σήμερα υπερασπίζονται των δικαιωμάτων αυτών. Ο λόγος στην ΙΕΔ παρακαλώ. Bonjour, merci, Ευχαριστώ πολύ και εμείς συμμεριζόμαστε την έκφραση αυτής της λύπης διότι δεν είναι παρούσε συγκεκριμένες προσωπικότητες εδώ. Θα ήθελα όμως να σταθώ στο θέμα της εξωτερικής πολιτικής και των σχέσεών μας με την Κούβα. Και ε, καταγράφω ένα σχόλιο ως προς την προγενέστερη αποτυχία μας Είχαμε μια στρατηγική εδώ και 20 χρόνια που δεν απέδωσε. Δηλαδή μιλήσαμε, είχαμε συνομιλίες, πολλές φορές δεν συμφωνούσαμε, αλλά θα δούμε από εδώ και στο εξής που θα φτάσουμε με το διάλογο αυτό. Πέρσι τον Οκτώβριο είχαμε το διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα που προβλέπεται από τον πολιτικό διάλογο και συνεργασία. Αυτός ο διάλογος ε, έγινε στις Βρυξέλλες. Ασχοληθήκαμε με πολλά θέματα, ακόμα και με αυτά που δεν μας βρήκαν σύμφωνους. Ένα ήταν ε, η βία, η βία κατά των γυναικών και η Κούβα αναγνώρισε ότι υφίσταται πρόβλημα και είπαμε ότι θα συνεργαστούμε για την αντιμετώπιση του. Είναι σαφές ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα αποτελεί αντικείμενο ε, δημόσιας θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι βρέως γνωστή. Η κοινωνία των πολιτών ε, είναι ε, σημαντικός συνομιλητής. Όπως ξέρετε υπάρχουν μηχανισμοί συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών. Γνωρίζουμε ότι πρόκειται για δύο παράλληλες ε, κοινωνίες των πολιτών, η επίσημη και η παράλληλη εμείς πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτόν τον διάλογο και με την παράλληλη κοινωνία των πολιτών, να έχουμε δηλαδή έναν διάλογο χωρίς αποκλισμούς ενός τμήματος της κοινωνίας των πολιτών. Είτε βρίσκεται στην Κούβα, είτε εδώ και γι' αυτό ενθαρρύνουμε το διάλογο που γίνεται σήμερα και αυτή τη βδομάδα, διότι θα έχουμε συνεργασία και αυτή τη βδομάδα με την διπλωματική αντιπροσωπεία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, λέει πρόεδρος και διακόπτη. Euh, avant de commencer le que Bernard Guetta souhaite euh, intervenir entre le Θα θέλατε ε, να λάβετε το λόγο για να συζητήσουμε το θέμα μεταξύ Κούβας και Τουρκίας. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να ενημερώσω την Επιτροπή μας για το γεγονός ότι ανέλαβα μία προσωπική πρωτοβουλία πέρα από οποιαδήποτε πολιτική ομάδα συμπεριλαμβανομένης και της δικής μου. Έγραψα λοιπόν στους προέδρους και τις προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να συνυπογράψουν και να δημοσιεύσουν μία δήλωση αλληλεγγύης και διαμαρτυρίας κατά του απαράδεκτου ε, και στη γυρού δράματος που γνωρίζουμε στη βορειοδυτική Συρία. Δεν πρόκειται για εκατοντάδες φυλακίσεις, πρόκειται για την τύχη εκατοντάδων χιλιάδων αμάχων ανδρών, γυναικών και παιδιών κάθε ηλικίας που βομβαρδίζονται συστηματικά εδώ και εβδομάδες που δυστυχώς ε, πλήττονται από το κρύο και λιμοκτονούν γιατί δεν υπάρχει τρόπος πια να λάβουν ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό γίνεται κάτω από τα ίδια μας τα μάτια και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση στον κόσμο η οποία ε, να διαμαρτυρηθεί. Κατανοούμε βεβαίως ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία αλλά και μία κόποση ε, έναντι του Συριακού δράματος. Αυτό εξηγεί και τις καθυστερήσεις ε, έκφρασης διαμαρτυρίας. Όμως το κοινοβούλιο μας δεν μπορεί να παραμείνει αδιάφορο και να μην αντιδράσει ενώπιον ενός τέτοιου δράματος. Θα πρέπει εμείς να κινήσουμε διαμαρτυρία και να εκφράσουμε την αγανάκτηση της διεθνούς κοινότητας. Γι' αυτό αυτό έστειλα επιστολή στους προέδρους των ομάδων, των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και απέστειλα επιστολή και στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου για να ζητήσω την υποστήριξη ως προς αυτό το διάβημα. Ήθελα να σας πληροφορήσω επ' αυτού και να σας πω ότι αυτό το έκανα πέρα από οποιαδήποτε πολιτική και ιδεολογική σκέψη. Ευχαριστούμε Μπερνάρ. Εγώ συμφωνώ απολύτως με την πρωτοβουλία που ανέλαβες και νομίζω ότι μπορούμε όλοι να διαβιβάσουμε το μήνυμα αυτό, το αίτημα αυτό για να υπάρξει μια θέση που θα αναλάβει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για το Μάρτιο έχουμε την προπαρασκευή της ε, συνάντησης ε, στην Τουρκία, της αποστολής στην Τουρκία, θα είναι το Μάρτιο. Είναι λοιπόν σημαντικό να μπορέσει να υπάρξει μια θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εν ώψη του Συμβουλίου που θα μπορούσε να εκφραστεί λίγο σαφέστερα σχετικά με την κατάσταση αυτή. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι. Θα καλέσω τώρα τους ομιλητές για την συζήτηση τη σχετική με την Τουρκία. Et donc on passe effectivement... Euh, Περνούμε λοιπόν σε αυτήν την ανταλλαγή απόψεων ε, επί της κατάστασης ε, στην οποία βρίσκονται οι καλλιτέχνες, ε, οι πανεπιστημιακοί, οι δικηγόροι στην Τουρκία σήμερα, σε συνέχεια του έργου που υλοποιεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είχαμε και έκτακτο ψήφισμα το Σεπτέμβριο πέρυσι και είχαμε προχωρήσει η ανταλλαγή απόψεων για την στρατιωτική επιχείρηση στη Βόρεια Συρία το Νοέμβριο. Ε, αναφέρομαι στην θλιβερή περίπτωση της δίκης Μπουγιού Καντά για τους εθελοντές ε, που κρίνονται ε, τρομοκράτες ως ε, μέλη τρομοκρατικής οργάνωσης. Δεν είναι η πρώτη φορά εξάλλου που τέτοιες κατηγορίες επιβάλλονται σε Τούρκους υπηκόους όταν αποκλίνουν από την γραμμή. Αύριο θα είναι η δίκη στην Κωνσταντινούπολη. 12 δικηγόροι ε, διακινδυνεύουν μέχρι και 15 χρόνια κάθερξης. Εμείς αποστήλαμε επιστολή στον εκπρόσωπο δικαιοσύνης Τουρκίας και στον κύριο Μπορέλ, ώστε η, η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορέσει να συμμετάσχει στην δικαστική ακρόαση αύριο. Έχουμε εδώ εκπροσώπους ε, της ε, μουσικής ομάδας Γιούχουν ε, για να μας εξηγήσουν την καταπίεση που υφίστανται εδώ και 10 χρόνια και άνω, κρατούνται, εχμαλωτίζονται, στην φυλακή υφίστανται βασανιστήρια, σωματικά και ψυχολογικά. Έχουν περιορισμό της ελευθερίας της εκφρασής τους παραβιάζεται κάθε διεθνές πρότυπο κράτησης ή φυλάκισης και αυτά θα τα διαβάσουμε στον Υπουργηγό Δικαιοσύνη στην Τουρκία. Έχουμε τους ακαδημαϊκούς, του πανεπιστημιακούς. Θυμίζω ότι το 2016 1118 ε, ακαδημαϊκοί και πανεπιστημιακοί υπέγραψαν μια επιστολή για την ειρήνη. Ε, όλοι αυτοί διώχθηκαν κάνοντας ε, τρομοκρατική προπαγάνδα. Η καταδίκη αυτή ήταν παραβίαση της ελευθερής έκφρασης ε, και θα έπρεπε να απελευθερωθούν όλοι οι συνυπογράφοντες της επιστολής αυτής. Ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να υλοποιηθούν οι ε, αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου στην Τουρκία όπως και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την απελευθέρωση του Οσμάν Καμπαλά που κρατείται εδώ και δύο χρόνια, να μην ξεχνούμε ε, του, τον εκπρόσωπο του ε, HDP και πρώην ε, υποψήφιο ε, για τις προεδρικές εκλογές σε Μίλντε έχουμε και τον ο Αρντογάν που απελευθερώθηκε μετά από τέσσερα χρόνια κάθεριξης σήμερα έχουμε τον κύριο Ισάν Σιμπελίκ, την κυρία Σιμπίλ Γκιοέ και τον κύριο Ερόλ Εντεργλού και τον κύριο Νευζά Τουσλού. Θα ξεκινήσω με την κυρία Σιμπιλ... Σιμπιλή. Ε, έχετε το λόγο για 10 λεπτά, παρακαλώ. Hepinizi selamlıyorum. Öncelikle Καλημέρα σε όλους. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ε, πρόσκληση που μου απευθύνατε για να μιλήσω για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ε, Τουρκία. Ε, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορώ να πω. Είναι δύσκολο να μιλήσω για αυτό το σημαντικό θέμα τόσο σύντομα. Η κυρία Πρόεδρος μίλησε για τα βασικά θέματα και θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια σημαντικά ζητήματα κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου. Αν υπάρχουν και άλλα ζητήματα, ευχαριστώ ε, να το δούμε μετά. Εγώ είμαι μέλος ε, της, ε, του γκρουπ του μουσικού ονόματι Eurum εδώ και 30 χρόνια. Εδώ και μία δεκαετία εδώ και 10 χρόνια ε, ζω στην Ευρώπη. Εξακολουθώ να είμαι μέλος του συγκροτήματος αυτού, συνεχίζω το έργο μου, το καλλιτεχνικό Οπότε τι συμβαίνει τώρα στην Τουρκία μετά από την απόπειρα πραξικοπήματος του 2015 αφού ε, κηρύχθηκε κατάσταση εκτακτής ανάγκης ε, αντιμετωπίσαμε διάφορες διώξεις και καταπίεση δεν μιλάμε όμως μόνο για καταστολή ε, έκτακτη αλλά και την τακτική θα έλεγα, την κανονική. Τι εννοούμε αυτό. Είναι μέρος της ε, καθημερινής μας ζωής στην Τουρκία. Όσοι ε, διαφωνούν, όσοι ψημένουν τα λάθη στην Τουρκία διώκονται και φημώνονται. Το σύστημα και η κεντρική κυβέρνηση πάντα δύο και τέτοιους ανθρώπους στην Τουρκία. Γι' αυτό είπα εγώ ότι πέρασα 10 χρόνια στην φυλακή. Τότε ακόμα μουσική έπαιζα, μουσικός ήμουν. Στήριζα εγώ και οι άλλοι διάφορους ακτιβιστές δύναμη συναυλίες Δεν μπορούσε να το απαγορεύσει αυτό η κυβέρνηση. Επειδή δεν μπορούσε λοιπόν να απαγορεύσει το καλλιτεχνικό μας έργο, άρχισε να λέει ότι είμαστε μέλη τρομοκρατικής οργάνωσης. Μας βασάνισαν, μας συνέλαβαν η κατάσταση άλλαξε από το πραξικόπημα και μετά. Πώς άλλαξε λοιπόν. Σήμερα ε, η κυβέρνηση ε, δεν προσπαθεί απλώς ε, να μας σταματήσει. Θέλει να μας φημώσει, θέλει να μας καταστρέψει εντελώς. τότε απλά ε, υπήρχε μία μαύρη λίστα στην παλαιά Τουρκία. Σήμερα πλέον απολύεται ο κόσμος. Αν, μιλήσει κάποιος, αν μιλούσε κάποιος καλλιτέχνης στο παρελθόν θα απαγορεύονταν οι συναυλίες τους. Τώρα όμως κλείνουν πολιτιστικά κέντρα για πολύ απλά πράγματα και ψευδείς ε, κατηγορίες. Ε, Φυλακίζεται το κόσμος για κανέναν απολύτως λόγο. Ο ο Τσελίκ ε, είναι σήμερα στην φυλακή. Στην φυλακή. Γιατί τραγούδισε ένα λαϊκό τραγούδι που είναι γνωστό στην Τουρκία εδώ και 45 χρόνια. Σεραλ Ακντά, επίσης μουσικός, ε, μέλος ε, του συγκροτήματος Μογγόλ. Βάλαν φυλακή γιατί τραγούδησε σε μια συναυλία. Κατηγορήθηκε, όπως ε, και ο άλλος φίλος, ως μέλος τρομοκρατικής οργάνωσης. Έξι μέλη του συγκροτήματός μας, του Γιουρούμ τώρα, είναι φυλακή. Κάποιοι άλλοι, όπως και εγώ, έχουμε περάσει από τις φυλακές. Έξι κρατούνται αυτή τη στιγμή. Και κατηγορούνται για τρομοκρατική προπαγάνδα και διάφορα τέτοια. Στον κινηματογράφο, λογοκρισία κάργα. Στα θέατρα επίσης. υπάλληλοι των κρατικών θεάτρων θεωρούνται δημόσιοι υπάλληλοι. Οι ηθοποιοί λέμε τώρα. Οι δημοσιογράφοι δεν μπορούν να μιλήσουν, δεν μπορούν να γράψουν ελεύθερα. Η κυβέρνηση προσπαθεί να εκπαιδεύσει, αν θέλετε, τους δικούς της. Αλλά διώκει και όσους ε, μιλάνε. Οπότε προσπαθούμε εμείς να αντισταθούμε. Κάποιοι προσπαθούν να βγάλουν κάποια κουβέντα να πούνε κάτι. Η αντίσταση αυτή συνεχίζεται. Όταν δεν φτάνει η αντίδραση προσπαθούμε να αντισταθούμε. Τώρα τα μέλη της ε, ομάδας μας ε, έχουν, πάει, έχουν περάσει απεργία πείνας. Και ζητάμε τέσσερα πράγματα. Ξεκίνησαν δε απεργία πείνας στις 16 Μαΐου 2019. Ορίστου διαρκείας. Και ε, ζητάμε κάποια πράγματα για να ευαισθητοποιήσουμε την διεθνή κοινότητα και έκτοτε λέμε το εξής. Δεν θέλουμε να κλείνουν ε, πολιτιστικά κέντρα, να γίνονται επιδρομές ε, όπως ε, και στο κέντρο του Γιουρουμ. Το πολιτικό μας ε, κέντρο υπέστη επιδρομές πάνω από 10 φορές. Έσπασαν τα μουσικά μας όργανα, ε, μας συνέλαβαν, έσκησαν τα βιβλία μας και διάφορα τέτοια. Την δέκατη δε φορά οι φίλοι μας που ήταν υποκράτηση, η συνελήφθησαν δεν ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Όλα δε τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος αναζητούνται. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ. Και τώρα με έχουν επικηρύξει. Δηλαδή αν με δώσουνε θα πληρωθούν οι άνθρωποι. Η μέλη μας τα, μέλη μας πάλι συνελήφθησαν πάλι πρόσφατα τα διάφορα πολιτιστικά μας κέντρα κλείνουν και διάφορα μέλη του συγκροτήματος μας συμμετείχαν στην απεργία πείνας τώρα ξεκίνησαν την απεργία θανάτου όπως λέμε είναι πάρα πολύ δύσκολο δεν θέλουν να πεθάνουν, αυτοί θέλουν απλά να είναι καλλιτέχνες. Και του λέμε, θα αντισταθούμε ακόμα και για σας που είστε ε, εχθρικοί. Γιατί ε, σήμερα καταπιέζουν εμάς, αύριο θα καταπιέσουν εσάς. Γι' αυτό αντιστακόμαστε. Βεβαίω. Ε, οι διώξεις είναι και άλλες πολιτικές λοιπά. Ο Μπρένγκοκτσέκ εξακολουθεί να είναι φυλακισμένος και στην τελευταία κρόαση δεν απελευθερώθηκε. Είναι τώρα στην 246η μέρα απεργίας πείνας. Τον Μάρτιο θα ξαναδικαστεί. Δεν ξέρω αν θα φτάσει μέχρι τον Μάρτιο αν Ελπίζω πραγματικά να μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε, να τον βοηθήσετε κι εσείς. Να βοηθήσετε την αντίσταση στην Τουρκία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ισάν για αυτή τη μαρτυρία σας, τη μαρτυρία από το Γιορούμ, καθώς και τους καλλιτέχνες που αντιστέκονται σήμερα. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Σιμπίλ Τζοέ που είναι δικηγόρος στη Λιέγη και επικεφαλής της ομάδας CHD Ευχαριστώ πολύ. Είμαι δικηγόρος, δικηγόρος στη Λιέγη και εκπροσωπώ Τούρκους ε, δικηγόρους που βρίσκονται στην Τουρκία ή στη Λιέγη. Παρακολούθησα αυτή τη ε, μαζική δίκη που έγινε και πολλές φορές δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει δίωξη και άλλων δικηγόρων αλλού. Γίνεται λόγος για ανεξαρτησία του δικαστικού τομέα και ελεύθερη εκπροσώπηση. Δυστυχώς όλοι αυτοί οι δικηγόροι διώκονται υπό την επωνυμία της τρομοκρατίας, ότι συμμετέχουν σε μία ε, τρομοκρατική οργάνωση και ο Μπαρ Κιμκί θεωρείται ότι είναι ο επικεφαλής. Αυτές οι κατηγορίες ε, δυστυχώς δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν με απόφαση του δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης και η φυλάκιση, η κάθυρξη είναι 18 ετών. Ακόμα και αν εφεσιδικήσουν δεν είναι σίγουρο ότι θα μειωθούν οι ποινές τους, οι ποινές των συνηγόρων αυτών. Οι συνήγοροι αυτοί υπερασπίζονται την ελευθερία λόγου και υπερασπίζονται πρόσωπα που έχουν βασανιστεί στις φυλακές και θεωρούνται ότι δυστυχώς, δυστυχώς συμμετέχουν σε τρομοκρατικές οργανώσεις. Πρόκειται για κατηγορίες ε, οι οποίες δεν έχουν βάση. Πολλές φορές οι καταγγελίες είναι ανώνυμες και πολλές φορές έχουμε μάρτυρες οι οποίοι πολλές φορές ε, προβαίνουν σε μαρτυρίες για να μειωθούν οι δικές τους πίνες και δεν ξέρουν καν για ποια δίκη καλούνται ως μάρτυρες. Διαπίστωσα ότι οι συνήγοροι υπεράσπισης δεν μπόρεσαν να μπουν στην αίθουσα στην διαδικασία επακροατηρίου. Αυτό αποτελεί βεβαίως ε, παραβίαση των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων. Το γεγονός δηλαδή ότι οι συνήγοροι υπεράσπισης διώκονται και εκδιώκονται από την αίθουσα. Μπροστά σε αυτές τις ιστοδυναικές δίκες, οι δικηγόροι έχουν προβεί σε απεργία πείνας από τις 3 Φεβρουαρίου, αλλά Μερικοί συμμετέχουν σε απεργία πείνας πάνω από 40 ημέρες και θα ήθελα να επισύρω την προσοχή σας ότι η επόμενη διαδικασία επακροατηρίου θα γίνει στις 4 Απριλίου και αφορά δύο δικηγόρους, την Βοιάσναν και η Ναϊτάι, που ε, διώκονται και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει μαζική παρουσία και ευρωβουλευτών, αν γίνεται. Η Ασλάν είχε ε, βασανιστεί και είχε χτυπηθεί κατά την κράτησή της και αυτό φάνηκε και από τα τραύματα που είδαμε στο πρόσωπό της όταν παρουσιάστηκε στη δίκη. Ζήτησε να γίνει μια πραγματογνωμοσύνη ως προς, τις, ε, ως προς τα χτυπήματα που δέχτηκε, δικαίωμα το οποίο της αρνήθηκαν. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο πίεσης έτσι ώστε να μην συνεχίζεται αυτή η σωματική και ψυχολογική βία. Επίσης, στην δίκη της 4ης Απριλίου θα πρέπει να παρευρεθούμε και να υποστηρίξουμε ε, μαζικά τους ε, κατηγορούμενους. Πρόκειται για μία δίκη η οποία ε, είχε ήδη αρχίσει από το Μάρτιο του 17 μέχρι το Μάρτιο 18 διακόπηκε και τώρα περιμένουμε την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου θα πρέπει να είμαστε παρόντες και να γνωρίζουμε τις εξελίξεις εκ του σύνεγγυ στην Τουρκία. Ως προς την ανεξαρτησία του δικαστικού τομέα στην Τουρκία, η κατάσταση είναι δυστυχώς τραγική. Μετά την απόπειρα πραξικοπήματος το Ιούλιο του 2006 έχουν απολυθεί 5.000 δικαστικοί υπάλληλοι. Πρόκειται για τεράστιο αριθμό. Έχουν αντικατασταθεί όλοι χωρίς να υπάρχει ε, εγγύηση αμεροληψίας που υποτίθεται συνοδεύει το δικαιοδοτικό. Επίσης το θέμα είναι πολύ λεπτό γιατί υπάρχει μεγάλη πίεση. Αρκεί ένας δικαστής να μην αποφασίσει όπως θέλει η εξουσία για να βρεθεί κατηγορούμενος, δηλαδή από τη μία πλευρά του εδωλίου στην άλλη. Αυτό είδαμε και στην περίπτωση του ε, συνήγορου Σετσλίκ Υπάρχει μεγάλη πίεση, πίεση στο δικαστικό τομέα. Ως προς τους συνήγορους έχουμε πάνω από χίλιους, 1500 που διώκονται μετά το 2016. Οι 600 έχουν φυλακιστεί και 384 έχουν καταδικαστεί σε 2.000 έτη φυλάκισης, καταλαβαίνετε. Γιατί μιλάμε, δηλαδή δεν τηρούνται οι διαδικασίες της Αβάνας και φημώνεται ο δικαστικός τομέας. Θα έπρεπε λοιπόν να γίνουν συστάσεις και εδώ μιλώ για την οργάνωση Lawyers for Lawyers. Έχουμε και εκπροσώπους εδώ. Πρόκειται για συστάσεις οι οποίες θα πρέπει να προωθηθούν προς την κυβέρνηση της ε, Τουρκίας. Θα πρέπει να σταματήσει η δίωξη των συνηγόρων να μην διώκονται με βάση την σύμβαση της Σαβάνας των Ηνωμένων Εθνών και η Τουρκία να δεχτεί την ε, ανεξαρτησία του δικαστικού τομέα, να μεταρρυθμίσει τους νόμους περί τρομοκρατίας που χρησιμοποιούν πολλά θεσμικά όργανα και τομείς να σταματήσουν τα βασανιστήρια κατά των συνηγόρων στις φυλακές και φυσικά να ασκήσουμε πίεση όλοι γιατί πρέπει να επαγρυπνούμε και φυσικά να είμαστε και αλληλέγγυοι προς τους συναδέλφους, αλλά διότι ποτέ δεν θα μπορούσαμε να αποφύγουμε ένα γενικότερο φήμοτρο του δικαιοδοτικού και μπορούν να γίνουν και πολλές ολιστήσεις στο μεταξύ. Σας ευχαριστούμε. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στους δημοσιογράφους, ε, εκπρόσωπο των ε, δημοσιογράφων χωρίς σύνορα, μιας οργάνωσης ε, στην Τουρκία συνδεμένος μαζί μας μέσω Skype που καλύπτει πολιτικά, πολιτιστικά και κοινωνικά ζητήματα, ιδιαίτερα τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχετε 10 λεπτά για να μας παρουσιάσετε την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία. Παρακαλώ. Can you hear me? Με ναι, ακούτε? Ναι. Κυρία Πρόεδρε, Αγαπητοί συμμετέχοντες, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση αυτή. Θα σας παρουσιάσω τους μουσιογράφους χωρίς ε, εκπροσωπό, τους μουσιογράφους χωρίς σύνορα ε, και παρακολουθώ τα θέματα ελευθερίας του τύπου εδώ και 25 χρόνια. Πηγαίνω δύο-τρεις φορές ε, την εβδομάδα στα δικαστήρια της Κωνσταντινούπολης και παρακολουθώ τις μαζικές δίκες κατά των δημοσιογράφων. Κοιτάξτε, ε, αυτό το οποίο στο παρελθόν ήταν ε, πρόβλημα του δικαστηρίου και της δικαιοσύνη. μετά το απόπειρα πραξιωμάτων του 2016 έγινε πλέον πιο συστημικό. Οι δημοσιογράφοι ε, είναι υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης υφίστανται πολιτικές πιέσεις και οι δημοσιογράφοι πιέζονται ε, για να προσαρμοστούν και να υφετήσουν έναν ε, πατριωτικό ας πούμε τρόπο ε, εξάσκησης του επαγγελματές τους. δεν είναι μόνο το 25% των ΜΜΕ που ελέγχεται αμέσως ή εμέσως, αλλά και οι υπόλοιποι σταθμοί και εφημερίδες υφίστανται δικαστική παρενόχληση και διοικητικά μέτρα. Ε, υπάρχουν ας πούμε οι λεγόμενες κάρτες τύπου, η διανομή των διαφημίσεων, αλλά και υπομορφή απαγόρευσης ε, του διαδικτύου με βάση την ε, διεύθυνση τη διαδικτυακή ή του περιεχομένου. Οπότε η κριτική πλέον ε, στα ΜΜΕ δεν είναι ευπρόσδεκτη και η κάλυψη μεγάλων ζητημάτων που σχετίζονται με την οικονομική κρίση, τα μέτρα ασφαλείας, τις πολιτικές ασφαλείας στην Συρία ή αλλού ή ζητήματα που αφορούν το Κυπριακό ή μεμονωμένη κριτική όλα αυτά είναι κάποια ζητήματα τα οποία θεωρούνται ταμπού στην ε, σύγχρονη Τουρκία. Λοιπόν, πρέπει επίσης να αναφέρουμε την αντιτρομοκρατική νομοθεσία γιατί έχει δημιουργήσει ακριβώς ε, μια αυτολογοκρισία στο τσατουρκικά τουρκικά μήμυε δεκάδες ε, εφημερίδες δικάζονται αυτή τη στιγμή είτε στην Κωνσταντινούπολη είτε στην Άγκυρα είτε στο Ντιγιαρμπακύρ. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το πολιτικό κλίμα μας σωθεί να πούμε ότι το πακέτο αυτό της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης που πέρασε τον Οκτώβριο δεν αρκεί για να αντιμετωπίσουμε αυτή την εχθρική παρέμβαση κατά των δημοσιογράφων στην Τουρκία. Δεν αρκεί απλά μια φράση που λέει ότι οποιαδήποτε κριτική δεν θα πρέπει να είναι αντικείμενο έρευνας ή ποινική δίωξης. Δεν θα τελειώσει έτσι αυτό αυτή η παρενόχληση όσο, παραδείγματος χάρη, το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο δεν είναι ανεξάρτητο. Όταν οι δικαστές ε, και οι εισαγγελείς αξιολογούνται με βάση τις αποφάσεις που βγάζουν ειδικά για πολύ ε, συμβολικές ε, δίκες ε, δημοσιογράφων όπως οι δίκες της Χουριέτ, του Σουσλοκ, η περίπτωση του Αχμέτ Αλτάν που παραμένει φυλακισμένος εδώ και τρία χρόνια. Μην ξεχνάμε αυτή η διακεκριμένοι δημοσιογράφοι καταδικάστηκαν επειδή υποστήριξαν μια παράνομη οργάνωση και τους κατηγόρησαν για συμμετοχή στην απόπειρα πραξικοπήματος. Ο Αχμεταλτάν καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκιση. Όμως εντός μιας εβδομάδας ε, από όταν διατάχθηκε η αποφυλάξη τους ξαναβρέθηκαν στη φυλακή γιατί ο εισαγγελέα Κωνσταντινούπολη άσκησε έφεση. Ας ε, δούμε ένα άλλο παράδειγμα, η περίπτωση της ε, Τζουμχουριέτ. Ε, το δικαστήριο απέριψε την άποψη του εφετίου και είπε ότι πρέπει να καταδικαστούν σε φυλάκιση επειδή στήριξαν ε, την οργάνωση ΦΕΤΟΕ του Γκιουλέν παρά το ότι ίσως ξέρετε ότι η γραμμή της Χουριέτ δεν έχει ούτε μία σχέση ε, με την οργάνωση αυτήν. Και τέλος, το τελευταίο παράδειγμα, οι δίκες της εφημερίδας Σιωτζιού μία από τις ε, κυριότερες ε, εφημερίδες που αντέδρασε κατά της ε, ενδυνάμωσης του κινήματος του Γκιουλέν εντός του κρατικού μηχανισμού και οι δημοσιογράφοι και οι αρχισυντάκτες αυτής της εφημερίδας ε, καταδικάστηκαν ε, πρόσφατα επίσης. Οπότε χωρίς ένα σύστημα ελέγχου της εξουσίας ε, στην Τουρκία χωρίς να σταματήσει η πολιτική παρέμβαση Ε, μπορείτε να περάσετε εσείς διαφορά. Ε, ε, μπορούν να περάσουν κάποιες αλλαγές που θα λένε ότι το ανώτατο δικαστήριο πλέον έχει αρμοδιότητες για την ελευθερία έκφρασης ή υπάρχει περιορισμός στην προφυλάκηση αλλά όσο υπάρχει ένας φορέας που υποτίθεται ότι ε, είναι αυτόνομος από τις ε, πολιτικές ε, πιέσεις. Η παρενόχληση των ΜΜΕ στην Τουρκία δεν θα τελειώσει δυστυχώς. Ένα παράδειγμα να σας δώσω. Είναι αυτό το θέμα των δημοσιογράφων που ασχολούνται με ζητήματα διαφθοράς, οικονομικής διαφθοράς. και τώρα αντιμετωπίζουν ε, πέντε χρόνια φυλάξη γιατί αναφέρονται στην υποτίμηση της ε, τουρκικής λίρας ε, πέρσι και οι δημοσιογράφοι του Bloomberg είναι μεταξύ των έξι δημοσιογράφων που αντιμετωπίζουν πιθανή ποινή πέντε ετών φυλάξης επειδή δυσφημούν την τουρκική οικονομία. Ένας άλλος δημοσιογράφος ε, αντιμετωπίζει πρόστιμο 150.000 ευρώ ε, επειδή άσκησε κριτική σε ατασταλίες ε, του οικονομικού συστήματος σε μεγάλους επιχειρηματίες που εμπλέκονται σε τραμπουκισμούς ή ζητήματα διαφθόρας πολλοί δημοσιογράφοι επίσης ε, που καλύπτουν τα Paradise Papers, ε, Panama Papers ε, κτλ. Έχουν επίσης διωχθεί τα τελευταία τρία χρόνια και καταδικαστεί επίσης. Όπως η περίπτωση Κιουλίνιν Κέρ, επειδή έναν δημοσιογράφο δηλαδή της Τζουμχουριέτ, η περίπτωση και πολλών άλλων δημοσιογράφων που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Το πρόβλημα λοιπόν που αντιμετωπίζει αντιμετωπίζουν τα ΜΜΕ στην ε, Τουρκία είναι πλέον συστημικό καθώς ε, τα θεσμικά όργανα που ρυθμίζουν το ζήτημα αυτό πλέον δεν είναι ανεξάρτητα αλλά δρούν εντός του προεδρικού συστήματος, ελέγχονται από ένα πολιτικό κύκλωμα εκατοντάδες δημοσιογράφοι αναμένουν ακόμα την έγκριση της κάρτας δημοσιογράφου. Και όλα αυτά καταλήγουν σε μια αυτολογοκρισία των δημοσιογράφων. Τα διοικητικά μέτρα είναι όλο και πιο διαδεδομένα. και δεν υπάρχει και κάποια διαδικασία προσφυγών δυστυχώς. Κατά την άποψη λοιπόν των δημοσιογράφων χωρίς ε, σύνορα θα θέλαμε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και το Συμβουλίο της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι πιο δυναμική όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της ε, δικαιοσύνης. και να δουν τις διαφορές πτυχές της ελευθερίας των ΜΜΕ στην διαδικασία αυτή. και είναι αυτό για εμάς ένας όρος εκ των όνου κάνευ. Όπως ε, παραδείγματος χάρη το άρθρο που αφορά την εξύβριση του Προέδρου ή την εξύβριση των δυνάμεων ασφαλείας και των οργάνων του κράτους, το άρθρο 41 που αφορά την ε, προσβολή ε, κατά λειτουργών του κράτους ε, και μελών της κυβερνήσεως το άρθρο 251 μια σειρά τροποποιήσεων που θέλουμε να δούμε για να σεβαστεί η Τουρκία τις ε, διεθνείς ε, δεσμεύσεις της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που μας είπατε. Και αντιλαμβάνομαι ότι είστε και εσείς ε, στο στόχαστρο επειδή μας μιλάτε σήμερα. Ελπίζω λοιπόν να πάνε όλα καλά στην Τουρκία. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Νευζάτος Λου, πρώην κοσμήτορ ε, του Πανεπιστημίου της ΣΥΦΑ. Θα μας παρουσιάσει τον ε, ακαδημαϊκό, την κατάσταση των ακαδημαϊκών σήμερα. Δεν είναι εδώ σήμερα μαζί μας, αλλά μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή του ε, θα έχουμε τη σύνδεση. Thank you very much. Uh, Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την δυνατότητα. Ονομάζομαι Νευζάτ Ουσλού, είμαι καρδιολόγος και αφού ολοκλήρωσα στον Πανεπιστήμιο του Μαρμαρά ε, εργάστηκα στο μεγαλύτερο καρδιολογικό κέντρο στην Τουρκία μετά στο νοσοκομείο Μερμεντάκ Ορσόη αν ακούσαμε καλά και μετά στο Ισμύρ στη Σμύρνη σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο που είναι γνωστό ως Πανεπιστήμιο Γκυλάν. Μετά την απόπειρα πραξικοπήματος χρειάστηκε να διαφύγω στην Ολλανδία γιατί στην Τουρκία επικρατούσαν ε, ριζοσπαστικές αντιλήψεις Έχω μία σύνοψη καταρχάς της παρουσίασης για το καθεστώς εκτάκτου ανάγκης και τα έκτακτα διατάγματα και μετά για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και τις παραβιάσεις των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελεύθερης μετακίνησης και θα ολοκληρώσω με, κάποιες, με κάποια συμπεράσματα και συστάσεις. Μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα τον Ιούλιο του 2016 η κυβέρνηση κήρυξε καθεστώς εκτάκτου ανάγκης υπό το οποίο ο επικεφαλής ε, της κυβέρνησης έχει απεριόριστη αρμοδιότητα να τροποποιήσει το Σύνταγμα και έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματα πολλών ανθρώπων που έχουν καταδικαστεί τρεις μήνες κάθε ρήξη ο καθένας αν καταλάβαμε καλά τον ομιλητή. Μετά την επιβολή του καθεστώτος εκτάκτου ανάγκης η κυβέρνηση άρχισε να κλείνει πανεπιστημιακά ιδρύματα που έχουν σχέση με το κίνημα Γκιουλέν 25 αν ακούσαμε καλά ε, τμήματα ιατρικής, ένα από τα οποία στο Ισμύρ πέντε πανεπιστημιακές σχολές και πάνω από 5.000 ιδιωτικά ιδρύματα. Επίσης άνω των χιλίων ενώσεων, 19 συνδικάτα και συνομοσπονδίες, όλα αυτά τα έκλεισε η κυβέρνηση συνολικά από τον Ιούλιο του 16 μέχρι τώρα άνω των 3.000 σχολεία και κοιτώνες έχουν κλείσει από την κυβέρνηση. Τώρα οι ακαδημαϊκοί οι οποίοι επηρεάστηκαν από αυτό το πρώτο βήμα κυρώσεων άνω των 2.000 απολύθηκαν από 96 διαφορετικά κρατικά πανεπιστήμια αν ακούσαμε καλά τον ομιλητή αυτό συνεχίζεται 5.000 συνολικά 200 και άνω. από 117 κρατικά πανεπιστήμια μέσω 6 ειδικών διαταγμάτων. Επίσης περίπου 3.000 ε, βοηθοί καθηγητές απολύθηκαν επίσης επίκουροι με συγχωρείτε, ε, αλλά βέβαια δεν απολύθηκαν μόνο ακαδημαϊκοί από, τα, από τις σχολές Γκιουλέν, αλλά και όλοι αυτοί που είχαν υπογράψει την ε, διακήρυξη ειρήνης. Οι 378 εκ των συνυπογραφόντων ακαδημαϊκοί υπέρ της ειρήνης έχασαν τη δουλειά τους, 265 βρίσκονται υποδίκη και εκατοντάδες άλλοι ερευνώνται, διώκονται. Επίσης, σχεδόν 65.000 φοιτητές, σπουδαστές, χρειάστηκε να αλλάξουν σχολή, πολλοί έχασαν ε, τις ε, υποτροφίες τους και αρκετοί από αυτούς συνελήφθησαν. και εκτός από τους Τούρκους σπουδαστές έχουμε και ξένους που έχουν υποστεί συνέπειες από όλα αυτά, επιστρέφουν στις χώρες τους χωρίς να έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών τους και οι, όσοι φοιτητέ παρακολουθούν σχολές γκουλέν στο εξωτερικό έχουν απαγορευτεί, έχει απαγορευτεί η εισοδός τους στη χώρα. επικρατεί μια κατάσταση κατά την οποία κανείς δεν μπορεί να εκφράσει την αποψή του χωρίς φόβο. Δεν υπάρχει ελευθερία έκφρασης και γνώμης. Αυτό δεν επηρεάζει μόνο τους ακαδημαϊκούς αλλά και τις οικογένειές τους και τους πολίτες. Δεν μπορούν να εγκαταλείψουν τη χώρα, έχουν ακυρωθεί, αποσυρθεί τα διαβατήριά τους πολλοί κρατούνται, πολλοί υφίστανται βασανιστήρια, και έχουν διαφύγει στην Ευρώπη σε διάφορες χώρες Ο αντίκτυπος όλων αυτών στην Τουρκία έχει γίνει μία μελέτη για την περίοδο Ιανουάριος έως Μάιος του 17 με την αντίστοιχη περίοδο και για το 16 η οποία δείχνει σοβαρότατη μείωση υποβολών μελετών ε, ερεύνης ιδιαίτερα σε θέματα κοινωνιολογικά και στην ιατρική. το κράτος θα πρέπει να επιστρέψει ε, όλα, όλες τις εγκαταστάσεις των πανεπιστημίων που έχει κλείσει των πανεπιστημίων και των υπολείπων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και θα πρέπει να σταματήσουν οι διώξεις κατά των ε, θεωρούμενων ή υπόπτων για τρομοκρατική δράση, οι οποίοι πρέπει να απελευθερωθούν. Το μέλλον της ακαδημαϊκής ελευθερίας στην Τουρκία είναι αβέβαιο, γιατί εξαρτάται από ένα δημοκρατικό περιβάλλον και επομένως το μέλλον των ακαδημαϊκών στην Τουρκία θα είναι συνδεμένο με το μέλλον της ίδιας της χώρας. Η κατάσταση είναι απογοητευτική και γίνεται και χειρότερη και σύμφωνα με τον Μάρκο Νίλσον η παραβίαση της ακαδημαϊκής ελευθερίας στην Τουρκία χρήζει σοβαρή σημασία από την διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα. Εγώ προσπαθώ να οικοδομήσω μια καινούργια ζωή στις κάτω χώρες και πολλοί συνάδελφοί μου υφίστανται βασανιστήρια στην Τουρκία αυτή τη στιγμή. Ε, αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, ε, λέει η Πρόεδρος. Θα δώσω τον λόγο στον Σεργέη που είναι υπεύθυνο της ε, μεικτής ε, Επιτροπής για την Τουρκία και στον Νάτσο. Σεργέη και Νάτσο λοιπόν. Well, if Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και τον ε, Νάτσο. Σας ευχαριστώ για αυτές τις συγκινητικές ε, μαρτυρίες. Απλά να σας πω ότι σήμερα ε, συνεχίζεται η δίκη κατά 15-16 ατόμων για την υπόθεση Καβάλα και άλλων ε, διαμαρτυριών στην πλατεία Γκαζή. Ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, εμβληματικό ζήτημα, γιατί δεν είναι θέμα τρομοκρατίας, η αφορά την κοινωνία των ε, πολιτών που προσπαθεί να ανατρέψει μια κυβέρνηση με διαδηλώσεις. Κάτι το οποίο παρακολουθούμε εκ του σύνεγγης ε, είχα πάει εγώ σε μια συνάντηση παραμονή Χριστουγέννων. Πρέπει λοιπόν ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λέμε ότι ε, οι μεταρρυθμίσεις που γίνονται για τη δικαιοσύνη δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. Προσπαθούμε να κάνουμε κάτι από αυτού. Βεβαίως ε, παρακολουθούμε τις δίκες, έχουμε τα διάφορα ψηφίσματα τα οποία εφαρμόζουμε ή ζητάμε πολλές φορές, αλλά παράδειγμα τους χάρη ο δεύτερος αντιπρόεδρος ε, Σλίμ Ντεμιρέλ πέρσι προσπαθούσε να πάει να παρατηρήσει μια δίκη η κυρία Ντεμιρέλ ε, για βομβιστική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη δεν την άφησαν να μπει στο δικαστήριο ε, δηλαδή δεν μπορούμε πλέον να μπούμε στα δικαστήρια κάποιοι από μας εξέδωσα μια δήλωση και μια διαμαρτυρία που προωθήθηκε και στην ε, πρεσβεία. Πρέπει να το ερευνήσουμε αυτό. Είναι βουλευτή. Ε, εντάξει μπορεί να είναι κανεί υπέρ ή κατά, αλλά είναι βουλευτή ε, και είναι στο Προεδρείο της Αντιπροσωπεία μας. Αυτό ήθελα να τονίσω ιδιαίτερος. Ε, κάτι το οποίο επίσης είναι σημαντικό όσον αφορά τις προσδοκίες των Τούρκων ε, εταίρων μας. Πρέπει να δούμε τον ορισμό της τρομοκρατίας. Η προσπάθεια επανορισμού που έγινε στην πρώτη ε, νομική μεταρρυθμίση δεν γίνεται. Δεν μπορεί να είναι όλοι τρομοκράτες. Δεν μπορεί μια ολόκληρη χώρα να αποτελείται από τρομοκράτες. Η ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και δικαιοσύνης έχει διαταραχθεί εντελώ. Πρέπει να μιλήσουμε για ανθρώπινα δικαιώματα και κράτους δικαίου και όσον αφορά τα θέματα ασφαλείας. Να μιλήσουμε επίσης για αλλαγή δικαστών, να έρθει μια νέα γενιά δικαστών. Για να ανατραπεί το όλο σκεπτικό. και ο συναλφός εδώ πέρα μάλλον συμφωνεί μαζί μου. Αυτό είναι βασικό πρόβλημα γιατί έτσι θα αλλάξει το σύστημα για πάντα. Δηλαδή να υπάρχει κάποιος ο οποίος ε, δεν θα έχει τόσο μεγάλη πείρα στο σύστημα. Πρέπει επίσης να εφαρμόζονται οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σύμφωνα με το τουρκικό σύνταγμα οι νόμοι στην Τουρκία πρέπει να ερμηνευτούν υπό το φως διεθνών υποχρεώσεων, ειδικά υποχρεώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ομολογία του ΕΔΑΔ. Αυτό το λέμε συνεχώς. Η Καβάλα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, Ντεμιρτά ένα άλλο. Έχουμε πολλές αποφάσεις πλέον. Και βεβαίω, αν υπάρχει βεβαίω και κάποια επαφή με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, είναι πάρα πολύ άργο στο να εκδώσει αποφάσεις και έχουμε πάρα πολλά θύματα που είναι στο έλεος των τουρκικών αρχών. Αυτά είναι κάποια από τα σημεία τα οποία θίγουμε εγώ και ο Νάτσο σε τακτική βάση με τους, τους ομολόγους μας και τους τα λέμε αλλά να πω και κάτι άλλο ως ε, πρόεδρος της τουρκικής αντιπροσωπείας. Αυτό το οποίο δεν πρέπει να κάνουμε είναι να εργαλειοποιήσουμε την κατάσταση η οποία είναι καταστροφική όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, γιατί ίσως θα αποθήσουμε την ε, Τουρκία για χρόνια, ίσως και για αιώνες. Δεν είναι αυτό το σωστό και νομίζω ότι οι παρόντες συμφωνούν. Εγώ είχα Πολλέ συζητήσει με εκπροσώπου τη κοινωνία των πολιτών και αυτούς που είναι στι φυλακέ και κινδυνεύουν και όλοι μου λένε μην σταματάτε. Μην σταματάτε την διαδικασία κάποιας ε, μακροπρόθεσμης ευρωπαϊκής προσέγγισης ε, με την Τουρκία γιατί αν μα εγκαταλείψετε τώρα δεν έχουμε καμία ελπίδα. Οπότε το θέμα δεν είναι μόνο η άσκηση κριτική στην τωρινή κυβέρνηση, αλλά το μέλλον της κοινωνίας και της κοινωνίας των πολιτών. Σα ευχαριστώ. Σεργέη, θα δώσω λόγο στον Νάτσο. Θα μιλήσω ε, ισπανικά για να μπορέσω να δώσω περισσότερες ε, αποχρώσεις στο λόγο μου. Εργάζομαι εδώ και χρόνια ε, για τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία και το γεγονός είναι, γεγονός είναι ότι δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση μετά την απόπειρα πραξικοπήματος. Ίσα ίσα το αντίθετο. Υπάρχει συγκεντρωτισμός του καθεστώτος, όλα περνάνε από το παλάτι όπως λέμε και αυτό που εννοούμε είναι τον πρόεδρο και την ε, κοντινή του εξουσία. Και δυστυχώς ε, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε έκφραση κοσμικής ε, εξουσίας. Έχει δυστυχώς επικρατήσει ο Ισλαμισμός και το Κοράνι αποκλειστικά σε κάθε μορφή έκφρασης. Δυστυχώς το πραξικόπημα είναι το μεγάλο άλοθη της κυβέρνησης, το οποίο, ε, πάνω στο οποίο δημιούργησε ένα αφήγημα η κυβέρνηση γύρω από την απόπειρα δηλαδή πραξικοπήματος και δεν επιτρέπει καμία κρίση και κριτική έναντι της ε, κυβέρνησης. Υπάρχουν 12.000 ονόματα γύρω από το πραξικόπημα. Ε, είναι τα ονόματα όλων αυτών που στη συνέχεια διόρισε η κυβέρνηση έτσι ώστε να απομακρύνει ε, όλες τις ευρωπαϊκές ελίτ μέσα σε εισαγωγικά. Και αυτό αφορά και την καταπολέμηση του γιουλενισμού. δηλαδή το άλοθη του πραξικοπήματος δεν επέτρεψε καμία κρίση ή επίκριση και περνάμε στα πανεπιστήμια, στους ακαδημαϊκούς και ούτω καθεξής. Με αυτό το συγκεκριμένο αφήγημα ε, μιλά η επικριση και περναμε στα πανεπιστημια στους ακαδημαικους και ουτω καθεξης με αυτο το συγκεκριμενο αφηγημα μιλα η κυβερνηση για ένα κράτος υπό πολιορκία, μιλώντας για τους Κούρδους, βίαιους ημί, τους γκιουλενιστές, τη συνωμοσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ και του Ευρωκοινοβουλίου που προστατεύει κάθε μορφή τρομοκρατίας, άρα δεν επιτρέπεται κριτικός λόγος. Ο κριτικός λόγος σημαίνει τρομοκρατία και βέβαια και η στρέβλωση της, εν, της έννοιας της τρομοκρατίας και της πολιτικής τρομοκρασίας. Δηλαδή, στην Τουρκία τα πάντα είναι τρομοκρατία. Αν ένας φοιτητής ε, ε, μεταφέρει ένα tweet, γράψει ένα tweet για το πόλεμο στη, Συρία, είναι τρομοκράτης. Εάν ένας δάσκαλος δουλεύει στη Μαλαισία και ήταν γιουλενιστής πριν από 15 χρόνια είναι τρομοκράτης. Όποιος ε, επικρίνει το στρατό είναι τρομοκράτης και όποιος, ε, ε, ε οποιοδήποτε χρησιμοποιήσει βία και στραφή ενός, ε, κατά ενός τρομοκράτη είναι τρομοκράτης. Όλα είναι εκδήλωση τρομοκρατίας. Εάν ο φοιτητή, ο οποίος γράφει ένα tweet είναι τρομοκράτης, τότε τι είναι όλοι οι άλλοι, πώς θα ποιήσει η Τουρκία την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ορισμένες κουρδικές οργανώσεις στη Συρία είναι ε, τρομοκράτες επειδή ένας ε, φοιτητής σχολίασε, σχολίασε την κατάσταση αυτών των κουρδικών ομάδων. Ε, δηλαδή, πρόκειται για μια διαδικασία, διαδικασία φήμοτρου. Δηλαδή, ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι διαμαρτυρόμενοι, οι διαδηλωτές του πάρκου Γκεζή προηγήθηκαν της απόπειρα πραξικοπήματος. Παρόλα αυτά και αυτοί τώρα θεωρούνται τρομοκράτες. Ε, μιλά λοιπόν η κυβέρνηση για μια κατάσταση πολιορκίας στην οποία ζει η χώρα. Τώρα έχουμε τη δίκη του Γκεζή, αύριο θα έχουμε τη δίκη της Μπουγιουκάδα. Εγώ έχω να σας παρακαλέσω το εξής. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία, αλλά ε, να μας δείξει τις δικαστικές αποφάσεις. Εάν ε, ο Γενικός εισαγγελέα ε, διώκει κάποιον που έχει κριτική σκέψη, ε, μην μιλάτε για ε, μεταρρυθμίσεις, μιλήστε μου για τις δικαστικές αποφάσεις, γιατί έτσι κρίνεται μία κυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα αυτή. Όλοι μας έχουμε την τάση να πούμε «Α, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δυστυχώς η Τουρκία δεν θα φτάσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ας σταματήσουμε τη διαδικασία προσχώρησης». Όταν εγώ προσπαθώ να βάλω ένα πρόσκομα σε αυτό το αφήγημα, σκέφτομαι τον ε, καβάλα, σκέφτομαι τους άλλους διοκόμενους, τους δικούς σας πελάτες, τους ε, πελάτες των συνηγόρων, διότι το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε το μοχλό της προσχώρησης. Εάν η Τουρκία πάψει να είναι υποψήφια χώρα, τότε δεν θα έχουμε και την δυνατότητα να υπερασπιστούμε το 60% του τουρκικού πληθυσμού που τάσεται υπέρ του ευρωπαϊκού προσανατολισμού. Όπως είπα στον Σεργέη, βεβαίως θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα επικριτικοί σε αυτή την κρατική παράνοια, έναντι οποιασδήποτε κριτικής σκέψης, αλλά δεν μπορούμε να στρέψουμε τα νότα προς ένα 60% του πληθυσμού που οι περισσότεροι είναι νέοι και είναι υπέρ της Ευρώπης, είναι συνήγοροι, είναι ακαδημαϊκοί και θα ήθελαν να τους υπερασπιστούμε και μπορούμε μόνο μέσω της διαδικασίας προσχώρησης, υποψήφιας χώρας προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο να ξέρετε ότι μπορείτε να βασιστείτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα θέλαμε και εσείς να περάσετε το μήνυμα ότι η διαδικασία δεν είναι να παρετηθούμε από τη μελλοντική προσχώρηση, ίσα ίσα θα πρέπει να την επιδιώξουμε για να μπορέσουμε να είμαστε παρεμβατικοί στα δρόμενα της Τουρκίας. Ιζαμπέλ, για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω θερμά όλους τους ε, ομιλητές ε, για τις παρουσιάσεις τους. Ε, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολουθεί πολύ προσεκτικά τα όσα σημαίνει στην Τουρκία. Εμείς ε, παγώσαμε τα κονδύλια που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την κυβέρνηση, χωρίς όμως να παγώσουμε τους σπόρους εκείνους που υποστηρίζουν την κοινωνία των πολιτών. Νομίζω ότι αυτό ήταν πολύ σημαντικό στα πλαίσια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό. Εάν ξανατοποθετηθείτε, ήθελα να μας πείτε πώς βλέπετε ότι εμείς μπορούμε απτά και συγκεκριμένα να βοηθήσουμε, γιατί εμένα δεν μου είναι πολύ σαφές. Θα είμαι πολύ σύντομη. Αλλά ήθελα να σημειώσω ότι έχουμε προβλέψει μία αποστολή στην Τουρκία χωρίς να ξέρουμε αν τελικά θα υπάρξει άδεια, έγκριση, ελπίζω να υπάρξει. Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θα ήταν καλό να τους δούμε. Ποιοι είναι αυτοί. Όλα αυτά που μας λέτε και όλα αυτά που γνωρίζουμε μας δείχνουν ότι η Τουρκία δεν θα πω απομακρύνεται από το κράτος δικαίου, αλλά ε, εν πάση περιπτώσει βρισκόμαστε σε μια de facto κατάσταση απουσίας κράτους δικαίου. Και θα ευχαριστήσω και τους προηγούμενους ομιλητές και τον ε, προλαλήσαντα σχετικά με το καθεστώς ε, υποψηφίου της Τουρκίας. Κάθε φορά που μιλούμε για σχέσεις με χώρες που δημιουργούν προβλήματα κράτους δικαίου και θεμελιωδών δικαιωμάτων αναφερόμαστε στο κατά πόσο ποιο πλαίσιο, ποια συμφωνία μαζί τους θα μπορούσε να μας επιτρέψει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, να ασκήσουμε την πίεσή μας. Από τότε που είναι υποψήφια η Τουρκία μέχρι σήμερα, πώς έχει κινηθεί η πρόοδός της ως προς το κράτος δικαίου. Θα μπορούσε κανείς να επιχειρηματολογήσει αντίστροφα ότι όλα αυτά τα χρόνια που είναι υποψήφια η Τουρκία έχει απομακρυνθεί ακόμα περισσότερο από τις αξίες μας. Και επομένως είναι αυτή η οδός που πρέπει να ακολουθήσουμε. Εγώ ξαναθέτω λοιπόν το ερώτημά μου ποια θα έπρεπε να είναι η θέση μας για το καθεστώς υποψηφίου χώρας. Και δεν είναι αυτό το καθεστώς που μας, ήγησε, που μας οδήγησε με συγχωρείτε εδώ που βρισκόμαστε, αλλά έχοντας αυτό το καθεστώς η χώρα αυτή έφτασε εδώ που έφτασε. Οπωσδήποτε δεν είναι εύκολη η απάντηση, αλλά ευχαριστώ όλους για τις προσπάθειές σας. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Ροντρίγκες ε, για το Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι βέβαιο όπως είπε και ο Νάτσο ότι η απόπειρα πραξικοπήματος ήταν πολύ σημαντικό σημείο καμπής αλλά ήδη από πριν είχαν αλλάξει τα πράγματα. Υπήρχε μια περίοδος κατά την οποία είχαμε ελπίδες ότι η Τουρκία προχωρούσε, ότι υπήρχε ένα άνοιγμα δημοκρατικό και δικαιωμάτων, το οποίο ανταποκρινόταν στην απέτηση πολύ μεγάλου μέρους της κοινωνίας. Επίσης είναι βέβαιο ότι το 2012 ήδη η Τουρκία εμφανιζόταν ε, ως μία από τις χώρες με τους περισσότερους ε, φυλακισμένους ε, δημοσιογράφους μετά και τις εκλογές του 2015 και ιδίω μετά την απόπειρα πραξιοποιήματος υπήρξε μια πολύ μεγάλη αντίδραση και καταπίεση κατά πολύ μεγάλου μέρους της κοινωνίας. Ακούσαμε την κατάσταση των δημοσιογράφων, των ακαδημαϊκών, αλλά έχουμε και κρατικούς λειτουργούς, υπαλλήλους, δημοσίους υπαλλήλους γραμματείς των Υπουργείων που απολύθηκαν, απομακρύνθηκαν, φυλακίστηκαν, ακυρώθηκαν διαβατήρια οικογενειών, συγγενών όλων αυτών των ανθρώπων, δηλαδή μια συλλογική καταπίεση. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν υπήρξε κανένα στοιχείο που θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει ικανοποιητικό. Και νομίζω, όπως είπε και η προηγούμενη συνάδελφος, ότι πραγματικά πρέπει να σκεφτούμε πολύ προσεκτικά τα πράγματα ως προς την ε, διαδικασία προσχώρησης της Τουρκίας ή του καθεστώτος υποψηφιότητός της. Είχαμε πάντα πολλά εμπόδια σε αυτή τη διαδικασία, αλλά ήταν παρόν, ένα στοιχείο παρόν, στην τουρκική και στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα και φαινόταν κάποτε ότι είχαμε ένα μοχλό πίεσης. Αλλά από ένα σημείο και μετά η τουρκική κυβέρνηση αφιερώθηκε σε άλλα πράγματα, αποφάσισε να εγκαταλείψει αυτήν την οδό, να γίνει περιφερειακή ηγέτιδα, ε, και η κατάσταση εσωτερική της κοινωνίας Τουρκίας επίσης ε, επιδεινώθηκε. Και πρέπει να κάνουμε σημαντική διάκριση μεταξύ της κοινωνίας της Τουρκίας, της μεγάλης της πλειοψηφίας, που καθόλου δεν έχει εγκαταλείψει το όραμα της προσχώρησης στην Ευρώπη. Ο κύριος Ντελαγκούε και μετά θα επανέλθω στους ε, ΕΛΚ ε, για να έχουν ακούσει όλες τις πολιτικές ομάδες. Εμείς ως Γκουε αλλά και ως ΑΚΕΛ, ως αριστερά από την Κύπρο που έχουμε υποφέρει πάρα πολύ και συνεχίζουμε να έχουμε προβλήματα με την Τουρκία θα θέλαμε μια Τουρκία διαφορετική. Μια Τουρκία δημοκρατική, μια Τουρκία που θα σέβεται το διεθνέ δίκαιο, το δίκαιο τη θάλασσα, που θα συμβάλλει στην επίλυση μια πολύ μεγάλη πληγή ενό άλλου του προβλήματο του Κυπριακού και που θα σεβόταν βέβαια και του ίδιου του πολίτε στην κοινωνία τη. Δεν έχουμε μπροστά μα μια τέτοια Τουρκία. Δεν μιλάμε καν για έλλειψη κράτου δικαίου. Μιλάμε για έναν Ισλαμοφασιστικό καθεστώ και είναι ντροπή για την ίδια την Ευρώπη να συνεχίζει να θεωρεί αυτήν την Τουρκία ω υποψήφια χώρα. Θέλετε να είμαστε απόλυτα ειλικρινεί. Πολλά από αυτά τα οποία ακούσαμε ακούγονται ως έβυχα λόγια για να χαϊδεύουν τα αυτιά μας. Η Ευρώπη αποδεικνύεται εντελώς ανίκανη να κάνει οτιδήποτε ουσιαστικό, πλήρως υποταγμένη και εγκλωβισμένη στις πολιτικές της, αλλά και σε ό,τι αφορά στο μεταναστευτικό, στις απειλές που ε, βγάζει απέναντί της η Τουρκία. Ούτε οι άλλε μεγάλε δυναμεί στην περιοχή, όπω αποδεικνύεται στη Συρία και στη Λιβύη, είναι έτοιμε ή ικανέ ή πρόθυμες να ταρακουνήσουν την Τουρκία, να την πάρουν από το αυτή. Αυτή τη στιγμή και ρωτώ και αυτούς που έχουν μιλήσει ως εισηγητέ, γιατί θεωρώ ότι η τελευταία ελπίδα για να ξαναβρει η Τουρκία το δρόμο τη, το δρόμο προς την πραγματική δημοκρατία, είναι η εσωτερική αντιπολίτευση. Είναι η, ίδια η τουρκική κοινωνία. Και με προβληματίζει πάρα πολύ εάν μέσα σε αυτόν το κλίμα της τρομοκρατίας που ασκείται εκ μέρους του κυρίου Ταγίπ Ερτογάν αν έχουν απομείνει δυνάμεις εντός της Τουρκίας που να παλέψουν πραγματικά. Πράγματι είναι 50-50 μοιρασμένη και εκλογικά η χώρα. Διερωτούμε πραγματικά, δεν ξέρω, διερωτούμε αν αυτόν το 50% καταγράφεται με συγκεκριμένους τρόπους, με συγκεκριμένες ενέργειες, εάν υπάρχουν αντιδράσεις, εάν ασκείται πίεση πάνω στο κατεστημένο του κυρίου Ερτογάν για να αλλάξουν κάποια πράγματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φούρλας και ο Βαντάλεν μετά. Ο, πρώτα και μετά ο κύριος Βαντάλεν. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους ε, φίλους από την Τουρκία που είχαν το θάρρος να είναι εδώ σήμερα μαζί μας και να μαρτυρήσουν όλα όσα έχουν πει και να τους ζητήσω και ένα συγγνώμη. Συγγνώμη διότι αυτά που είπατε μπορεί να μεταφραστούν σε έναν ψήφισμα, σε μια ωρεολογία από μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να σα συμπαρασταθούμε φραστικά, α πούμε πολύ ωραία πράγματα, αλλά επί τη ουσίας δεν θα λάβετε τίποτα από εμά. Ξέρετε γιατί. Το είπαν εδώ και ακούστηκε και έχουν δίκιο συνάδελφοι. Η Τουρκία είναι υπό ένταξη κράτος μέλος και αυτός ο μοχλό πίεσης που θα έπρεπε να είναι για την Τουρκία είναι μοχλό πίεση για την Ευρώπη. Σε βάρο τη Ευρώπη. Τόσα χρόνια που είναι υπό ένταξη κράτο η Τουρκία, πέστε μου ποια διαφορά αν έχει σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε επίπεδο δημοκρατία. Ένα παράδειγμα να μου πείτε, μόνο που βοήθησε αυτή την ταξική πορεία. Θα μου πείτε τι εισηγήσε εκεί που πονάει η Τουρκία, που είναι η χρηματοδότηση. Διότι θα φύγετε από εδώ, μα είπετε αυτά που μα είπατε, μα είπετε πόσο κινδυνεύετε ότι οι άνθρωποι πάνε στη φυλακή διότι λένε ένα τραγούδι το οποίο δεν εγκρίνει το καθεστώ. Και εμεί εδώ θα πούμε πολύ όμορφα λόγια, αλλά θα συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε την Τουρκία. Αυτή είναι η Ευρώπη. Και αυτό το πράγμα, όσο δεν αλλάζει, δεν θα αλλάξει τίποτε. Και θέλαμε απολύτω έντιμο μαζί σα. Και δεν μιλώ ω Κύπριο, που είναι υποκατοχήν η πατρίδα του, μιλώ ω ένα Ευρωπαίο πολίτη, ο οποίο βλέπει αυτά που βλέπει έτσι το Ευρωκοινοβούλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα σας ε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ όσους ήρθαν σήμερα και μας μίλησαν. Ε, εκτιμούμε ιδιαιτέρως ε, το ότι διατρέχετε κίνδυνο για να μας μιλήσετε Πριν από μερικά χρόνια έκανα ένα μεγάλο ταξίδι και στην ε, Τουρκία σε διάφορες πόλεις ε, όπως ε, το Νίριατ και σε άλλα μέρη σε εκείνη την περιοχή και η κυβέρνηση Ερντογάν τότε το 2012 ήταν απασχολημένη με το να πατάσει τους αντιπάλους μεταξύ των οποίων και εκκλησίες και μονές ε, ε, από τους οποίους απαλωτριωνόταν ε, η ιδιοκτησία τους. Έχουν αποδεκτικά χαρτιά που πηγαίνουν στο 400 μετά Χριστού που αποδεικνύουν την συνεχή ιδιοκτησία τους. Λοιπόν, μετά από τέσσερις μήνες ε, δεχτήκαμε και τον ε, Παστορά Μπράνσον εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο οποίος είχε κατηγορηθεί επίσης για τρομοκρατία, όπως κατηγορούνται πανεπιστημιακοί, δημοσιογράφοι και δικηγόροι. Και έρχομαι στην ερώτησή μου. Η Ευρώπη εδώ και χρόνια ασχολείται με το θέμα της ένταξης της ε, Τουρκίας αλλά υπάρχει και μια διαφορετική κατεύθυνση. Ο Ερντογάν απομακρύνεται από την Ευρώπη, γελάει με την Ευρώπη, κουνάει το δάχτυλο στην Ευρώπη και η κατάσταση χειροτερεύει συνεχώς. Οπότε για εμένα το ερώτημα είναι τι θεωρείτε ότι πρέπει να κάνουμε στις σχέσεις μας με την Τουρκία. Σας ευχαριστώ. τον λόγο στον τον κύριο Νταμ ε, που εκπροσωπεί το Human Rights Watch και μετά θα σας δώσω λίγα λεπτά για να απαντήσετε σε κάποιες ερωτήσεις που υπευλήθησαν. Ο κύριος Νταμ. Ευχαριστώ που μας ε, προσκαλέσατε. Η διευθύντρια της ε, Τουρκίας παρακολουθεί διάφορες δίκες που διεξάγονται αυτήν την στιγμή θα ήθελα να επισημάνω μια άλλη κατηγορία ατόμων που υφίστανται διώξεις στην χώρα τους ε, δημάρχους ε, στην νοτιοανατολική Τουρκία. Οι αρχές ε, έχουν εντείνει τις διώξεις τους και στη μεθορική περιοχή με την Συρία καθερούν εκλεγμένους δημάρχους. Αυτή τη στιγμή 23 δήμαρχοι ε, είναι υποκράτηση με κατηγορίες τρομοκρατίας και στις 10 Φεβρουαρίου ένα δικαστήριο ε, φυλάκισε τον δήμαρχο του Ντιγερμπακύρ. Θεωρούμε ότι η κατάσταση θα συνεχιστεί και θα καταπατούνται τα δικαιώματα των πολιτών αλλά και των 8 εκατομμυρίων ε, πολιτών που τους εξέλεξαν. Αναφέρατε πριν το ότι οι τουρκικές αρχές δεν εφάρμοσαν την απόφαση του ΔΕΚ του 2018 για τον Ντεμιρτάς και έχουν μπει στο στόχαστρο και άλλοι αντιπολιτευόμενοι. Έχουμε πει στον Οσμάν Καβαλάν και άλλους για τους οποίους ο εισαγγελέα συζητάει η ε, για τρεις από αυτούς. Αυτό μας υπενθυμίζει το πώς έχει η κατάσταση και Βεβαίω παρά την δήλωση της εκπροσώπου της Κομισιόν και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης ε, που λένε ότι δεν είναι κατάλληλη η στιγμή ε, για να τα αναλάβει αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να μιλήσουμε για τους συμβαστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων που φυλακίζονται στην ε, Τουρκία ειδικά καθώς ε, σήμερα και πάλι αγνοήθηκε η απόφαση του ΔΕΚ από τα τουρκικά δικαστήρια. Λοιπόν, οι υποθέσεις αυτές ε, είναι απλά η κορφή του παγόβουνου. Χιλιάδες ε, άτομα έχουν διωχθεί με αστήρικτες κατηγορίες και φέδρες καταδίκης λοιπόν δεν θα πρέπει να μας παραπλανούν ε, οι υποσχέσεις για σχέδια μεταρρυθμίσεων. Θα πρέπει να δούμε τις εξελίξεις, τις διάφορες υποθέσεις που εκδικάζονται. Θα πρέπει ακριβώς ε, να επιδειχθεί η πολιτική βούληση για να σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα και να διασφαλιστεί μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη χωρίς ε, παρενόχληση. Και θέλουμε όλα τα θεσμικά όργανα να ε, πιέσουν την Τουρκία για να γίνει αυτό. Σας ευχαριστώ. Όστια. Έχετε το λόγο για ένα λεπτό και θα δώσω το λόγο στην ΕΕΔ για να απαντήσω στην ερώτησή σας τι μπορούμε να κάνουμε. Νομίζω ότι η παρουσία στη δίκη είναι σκόπιμη διότι περιορίζεται η εκδήλωση βίας και μπορούμε να λογοδοτήσουμε και ενώπιον διεθνών δικαστηρίων όπως του ΕΔΑΔ. Έχει μεγάλη σημασία για την στήριξη των πολιτικών κρατουμένων και για να κρίνουμε και τους δικαστές που είναι υπέρ της καταστολής, όπως του Ακάν Κυρλέκ. Να τον ρωτήσουμε γιατί ακριβώς, να του θέσουμε ερωτήσεις για τη στάση του. Δεν μπορώ να μιλήσω για τη διαδικασία προσχώρησης, ακούω τις παρατηρήσεις, να μην σταματήσουμε το διάλογο, Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει φτάσει σε μια συμφωνία με την Τουρκία για τους πρόσφυγες που δεν ευεργετεί κανέναν. Απλώς χρηματοδοτεί με κολοσιαία ποσά την τουρκική κυβέρνηση και δυστυχώς οδηγεί την ε, Ευρώπη σε πλήρη κατάργηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων γιατί φτιάχνουμε καταβλισμούς όπου ζουν άνθρωποι υπό απάνθρωπες συνθήκες. Θα πρέπει να ε, ασκήσουμε πίεση εκεί που μπορούμε δηλαδή. Θα ήθελα και εγώ να ε, εκφράσω τις ευχαριστίες μου και την ευγνωμοσύνη μου σε όλους τους συναδέλφους που συνέδραμαν σε αυτή τη συζήτηση, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ σε μία πρόταση που, στην οποία αναφέρθηκε ο Κύπριος Ευρωβουλευτής. Η πραγματική ελπίδα είναι οι άνθρωποι που ζουν μέσα στη χώρα, στην Τουρκία, που θα ταχθούν υπέρ της δημοκρατίας και της αντίστασης. Συμφωνώ μαζί σας. Τώρα, ως προς την αποστολή που θα ε, επισκεφθεί την Τουρκία και ποιοι θα πρέπει να είναι οι συνομιλητές. Ε, έχουμε ανθρώπους όπως την ε, Χελίν Μπερέκ, τον Ιμπραήμ Γκέτσεκ, οι οποίοι κάνουν απεργία πείνας, απεργία πείνας και βρίσκονται σε τελικό στάδιο. Επίσης θα πρέπει να επισκεφθείτε την νοτιοανατολική Τουρκία. Επισκεφθείτε φυλακές. Μπορούμε να σας δώσουμε ένα κατάλογο φυλακισμένων που θα μπορούσατε να επισκεφθείτε. Έτσι θα μπορέσετε να επηρεάσετε τα πράγματα γιατί αυτό θα δείξει στις εθνικές αρχές ότι κάνετε κάτι, αλλά οι δημοκρατικές δυνάμεις στη χώρα είναι η λύση. Έρολ, έχεις το λόγο αν θέλεις να πεις κάτι. Ναι, Πρόεδρε, ήθελα να επανέλθω στο ζήτημα του κατά πόσον υπάρχει ένα κίνημα αντίστασης στην Τουρκία. Αναφερθήκαμε σε διάφορα προβλήματα αλλά παρά την καταπίεση διάφορα κομμάτια της τουρκικής κοινωνίας και διάφορες ενώσεις μεταξύ άλλων και δημοσιογραφικές οργανώσεις ακόμα καταφέρνουν, προσπαθούν εν πάση περιπτώσει να, ενημερίσουν, να ενημερώνουν την κοινή γνώμη. Ε, και μετά τις ε, περισσινές εκλογές αναπτύσσεται ένα νέο ρεύμα ε, στην τουρκική κοινωνία τα, ούτως ή άλλως τα μέσα ενημέρωσης, τα επίσημα είναι ε, απλώς ε, φερέφωνα της κυβέρνησης μεταφέρουν την κρατική γραμμή και τίποτε άλλο και επομένως έχουν χάσει την αξιοπιστία τους. Υπάρχουν καινούργιοι τρόποι ενημέρωσης, υπάρχουν εναλλακτικά μέσα αλλά βεβαίω ε, η κυβέρνηση έχει αναλάβει και μέτρα περιορισμού του διαδικτύου, των συνδέσεων στο ίντερνετ και του περιεχομένου. Παρακολουθούμε την περίπτωση του Οσμάν Καμπάλα και ε, Μπούκαντα, Γκέζι επίσης και άλλες δίκες Νομίζω ότι οι σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας δεν θα πρέπει να γίνονται κατά τρόπον ηθικού διδάγματος ή επιβολής από τη μία πλευρά στην άλλη. Ε, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα που υπάρχει. Γιατί όποιο και να είναι το μέλλον, πάντα θα χρειαστεί να έχουμε στενές σχέσεις η Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, άνω των 5 εκατομμυρίων Τούρκοι διαμένουν, κατοικούν στην Ευρώπη, υπάρχει τεράστια κοινωνική και εμπορική διάδραση μεταξύ Τουρκίας και Ευρώπης. Και βεβαίως πρέπει να επικρίνουμε την κυβέρνηση. Αλλά οι θρησκευτικές τάσεις κάποιου κομματιού της κοινωνίας δεν είναι αναγκαστικά αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος κοινικού διότι και οι τοπικές πρόσφατες εκλογές έχουν δείξει ένα, ένα τοπίο αρκετά κινητικό, δυναμικό. Και ας δούμε αυτή τη δυναμικότητα ως ευκαιρία στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα μπορεί να επηρεάσει κάπως τα πράγματα. Ευχαριστώ, Ερόλ Διακόπτη Πρόεδρος. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Ο κύριος Νευζάτ έχει επίσης ένα λεπτό, αλλά ένα λεπτό και μόνο, γιατί πρέπει να δώσω το λόγο στην Επιτροπή και στην ΙΕΔ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα, θα μιλήσω και εγώ στα τουρκικά. Η κυβέρνηση Ερντογάν ε, προσπαθεί να υποσκάπτει μάλλον κάθε θεσμό στην Τουρκία. Τα πράγματα έχουν χειροτερέψει πολύ προκειμένου να ενισχύσουμε τη δημοκρατία στην Τουρκία πρέπει να κάνουμε ο καθένας ό,τι καλύτερο μπορεί. Δεν πρέπει να ξεχνούμε τους ε, φυλακισμένους ακαδημαϊκούς. Με αυτό θα ήθελα να κλείσω, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Ο λόγος τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ακολούθω στην ΕΕΔ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κοιτάξτε, η διάγνωση σημερινή δεν είναι καινούρια. Ε, λυπούμε. Διότι η Κομισιόν εδώ και χρόνια στην ετήσια έκθεσή της ε, διαπιστώνει την δυσάρεστη, την λυπηρή κατάσταση ε, του κράτους δικαίου μεταξύ άλλων που επικρατεί στην Τουρκία, την ελευθερία έκφρασης τύπου, δικαιοσύνης, τι όλο και μειούμενες ελευθερίες ε, για την κοινωνία των πολιτών, όλα αυτά έχουν ε, περιγραφεί συγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και στα πλαίσια του διαλόγου με την Τουρκία ακριβώς θα πρέπει να εστιαστούμε πιστεύω στην ερμηνεία, στον ορισμό τις τρομοκρατική δραστηριότητα ε, που υφίσταται, που χρησιμοποιεί η τουρκική κυβέρνηση και που είναι ευρύτατη. Εμείς εδώ και κάποια χρόνια κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε ε, οι ομόλογοι μας στην Τουρκία να συνεχίζουν μαζί μας ένα διάλογο για το κράτος δικαίου, για την ελευθερία έκφρασης και τύπου, για τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης για την προετοιμασία ενός νέου σχεδίου δράσεως για τα, δικαιώματα, για τα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά βεβαίως αντιλαμβανόμαστε και τους περιορισμούς του διαλόγου αυτού. Έχουμε κινητοποιήσει και τα μέσα που έχουν διαθεσή μας ε, βοήθειας, βοήθειας των ανεξάρτητων φορέων των κοινωνικών. Έχουμε αυξήσει τα κονδύλια που απευθύνονται στην ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών, τους υπερασπιστές ε, των δικαιωμάτων, τις ε, οργανώσεις ε, των εναλλακτικών μέσων ενημέρωσης, των ενώσεων ακαδημαϊκών και πανεπιστημιακών, με τους οποίους έχουμε υποστηρίξει ε, με ανθρωπιστική βοήθεια πολύ σημαντική μετά την απολυσή τους, πέραν της χρηματικής αυτής στήριξης, έχουμε 30 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για την κοινωνία των πολιτών που τα διαχειρίζεται πλέον η Επιτροπή και όχι οι τουρκικές αρχές. Ε, έχουμε ένα πρόγραμμα παρατήρησης ε, των ε, δικαστικών διαδικασιών που εξελίσσονται, ιδιαίτερα της περίπτωσης Γκεζή. Υπάρχει ένα συντονισμός στην Άκυρα μεταξύ των κρατών μελών για να παρακολουθούμε ακριβώς τις διαδικασίες αυτές και τις νομικές εξελίξεις εν γέννη. Διατηρούμε το διάλογο με τις τουρκικές αρχές και στα πλαίσια των επομένων συστάσεων του Συμβουλίου ελπίζουμε και το Συμβούλιο να προσθέσει την ενθάρρυνσή του προς τις τουρκικές αρχές ε, να, σέβονται, να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Η Εύα έχει το λόγο. For, for this. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι Εντάχει μπορώ να πω ότι η Επιτροπή παρουσίασε πράγματα που μας βρίσκουν σύμφωνους ε, και ιδιαίτερα οι επικρίσεις που αναφέρθηκαν από τους προσκεκλημένους μας ή από τους ευρωβουλευτές. Ε, όλα αυτά τα έχουμε αναγνωρίσει, η απο τους ευρωβουλευτες ολα ύπατη εκπρόσωπος, ο νυν ύπατος εκπρόσωπος, ε, γνωρίζουμε την κατάσταση στην Τουρκία και γνωρίζουμε ότι ε, συρρυκνούνται τα δικαιώματα. Δυστυχώς ακτιβιστές, ακαδημαϊκοί, ε, πολιτικοί σε εκλεγμένοι δήμαρχοι, όλοι αυτοί φυλακίζονται. Βλέπουμε λοιπόν ότι στο διάλογο μας με την Άγκυρα μπορούμε να πλαισιώσουμε σωστά τις ανησυχίες μας και να παρουσιάσουμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας ως προς την Τουρκία ως υποψήφια χώρα και ως μέλος, μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης. Θα πρέπει να τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα και η στρατηγική της υποψήφιας χώρας έχει προαναφερθεί. προαναφερθεί. Θα πρέπει όμως να φτάσουμε σε απτά μέτρα για να δούμε πως η έκβαση των δικαστικών αποφάσεων του Στρασβούργου εφαρμόζονται στην Άγκυρα ή αλλού στην Τουρκία. Κατά πόσο αντικατοπτρίζεται η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Τουρκία επίσης. Διαθέτουμε έναν μηχανισμό για την παρατήρηση των δικών. Ε, εμείς θα παρακολουθήσουμε τις ε, δύο δίκες αυτής εβδομάδας, Καβάλα και Γκεζή, και γίνεται αποτίμηση της κατάστασης σε τακτά χρονικά διαστήματα σε μια ομάδα εργασίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και εκεί συμμετέχουν και ΜΚΟ και οργανώσεις ε, κοινωνικής δικτύωσης και κοινωνίας των πολιτών. Επίσης, η αντιπροσωπεία μας ε, οργανώνει επισκέψεις σε ΜΚΟ ή πρόσωπα σε κίνδυνο, αντιρρησίες και ούτω καθεξής. Ε, τέλος, θεωρούμε ότι και στο Συμβούλιο της Ευρώπης πρέπει να θίγονται αυτά τα ζητήματα και εμείς ε, ήδη πέρσι αναφερθήκαμε στην Τουρκία τρεις φορές. Έχουμε όλα αυτά τα μέσα για να μπορέσουμε να ασκήσουμε πίεση σε μια υποψήφια χώρα. Σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση που ήταν ιδιαίτερα πλούσια. Σας ευχαριστώ για τις μαρτυρίες σας. Ελπίζω και προτείνω ως πρόεδρος να προβάλλουμε ένα ανακοινοθέν για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και αυτό αφορά και τον Νάτσο που είναι ο μόνιμος εκπρόσωπός μας στις σχέσεις με την Τουρκία. Θα σας προτείνω ένα κείμενο και θα μιλήσουμε και για τη σύσταση μίας αντιπροσωπείας η οποία θα είναι παρούσα στις δίκες και θα λάβει υπόψη τις συστάσεις των παρεμβενόντων. Μία αντιπροσωπεία ΑΦΕΤ θα μεταβεί στην Τουρκία την επόμενη εβδομάδα και ελπίζουμε να φυγούν παρεμφερή ζητήματα και έχουμε και μία αποστολή 3 με 6 Απριλίου, όπου βεβαίως θα λάβουμε υπόψη τις συστάσεις σας. Στα πλαίσια της συζήτησης μιλήσαμε και για το διάλογο με την Τουρκία ως υποψήφια χώρα και όλες τις απαιτήσεις και προαπαιτούμενα που μπορούμε να προβάλλουμε. Αυτό αφορά και την Τελωνιακή Ένωση, την οποία μπορούμε να προβάλλουμε ως οικονομικό μέσο μόχλευσης. Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε και τέτοια μέσα τα οποία να τα υποτάσσουμε στην τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί είναι ένας μοχλός ο οποίος δεν χρησιμοποιείται αρκούντος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ για τις μαρτυρίες σας και ευχαριστώ και τους καλεσμένους μέσω Skype. Σας ενθαρρύνουμε να συνεχίσετε την εξαιρετική σας εργασία. On va passer Τώρα περνάμε και κλεισμένων των θυρών, στη συνάντησή μας και κλεισμένων των θυρών, αλλά θα σας παρακαλούσα να αποχωρήσετε σύντομα.